με ιδιαίτερη χαρά να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση όλοι μαζί της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών. Σήμερα θα ασχοληθούμε απλώς και μόνο με την αναθεώρηση της οδηγίας των καθυστερήσεων πληρωμών. Προηγουμένως απλώς θα σας ζητήσω να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Είχαμε μια Εν μέρη συνάντηση των ε, συντονιστών σήμερα το πρωί θα συνεχιστεί και το απόγευμα. Θα σας ενημερώσω για τις αποφάσεις των συντονιστών αύριο το πρωί. Επίσης πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεών μας. 28 και 29 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου. Υποθέτω ότι συμφωνείτε. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε στις πρωινές μας εργασίες. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τους σκληρά εργαζόμενους, τη σκληρά εργαζόμενη μας, την Μπαρμπαρα Βάιλερ, που κάθεται δίπλα μου, για το έργο της σε αυτό το σημείο. Το ντοσιέ και να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπαλντασάρη που είναι ο συγητής της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων ο οποίος θα μας ενημερώσει για την ενισχυμένη συνεργασία. Είναι μεγάλη μας χάρη να σας έχουμε σήμερα εδώ κύριε Μπαλντασάρε θα μας πείτε και εσείς τις απόψεις και θα συμμετάσχετε στην ακρόαση. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που έχουμε διακεκριμένους ειδικού σήμερα μαζί μας. Τα βλέπετε στο πρόγραμμά σας, θα τους ε, παρουσιάσουμε εν καιρό μόλις περάσουμε στο, στην ακρόαση αυτή καθεαυτή. Να ευχαριστήσω και την κυρία Μπρίκμαν, την εκπρόσωπο της Επιτροπής, να τι εκεί είναι. Δεν ξέρω γιατί είσαστε τόσο μακριά από τους υπόλοιπους ειδικού. Ξέρω ότι η κυρία Λεμπάη ήταν απασχολημένη σήμερα παρόλο που ήθελε να είναι εδώ, την Γενική σας Διεύθυνση. Αλλά είναι χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας αφού παρακολουθείτε την εξέλιξη του ντουσιέ αυτού. Θα παρουσιάσετε τη μελέτη αντικτύπου. Από ό,τι ξέρω. Η γραμματεία μας ενημερώνει ότι έχουμε τον εισηγητή και της Επιτροπής Βιομηχανίας του κύριο Ντεάντζελης μαζί μας. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον δοσχέ αυτό και από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Η ακρόαση σήμερα έχει σκοπό να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία και προτάσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ειδικού και να δώσει συνέχεια στην, στο έργο της Επιτροπής μας καθώς επεξεργάζεται αυτή την πολύ σημαντική πρόταση. Ελπίζουμε λοιπόν ότι σήμερα το πρωί θα επιτελέσουμε πρόοδο. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να καλέσω τον, την εισηγητριά μας, την κυρία Βάιλερ, να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή και να παρουσιάσει και το έγγραφο εργασίας που έχει ετοιμάσει σε εσάς έγγραφο το οποίο κανονικά διατίθεται σε όλους, υπάρχει αντίτυπο λογικά και μετάφραση σε κάθε γλώσσα. Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είπατε με ιδιαίτερη ευγένεια ότι η ακρόαση αυτή σκοπό έχει να μας δώσει την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις των ειδικών και αυτές που είναι ειδικά σημαντικές για εμάς για να λάβουμε την απόφαση μας ως βουλευτές αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να γίνει πιο ουσιαστική η συζήτηση γιατί άκουσα εγώ κάποια πράγματα στα ΜΜΕ που θέλουν εδώ πέρα πως, ε, ότι θέμε εδώ πέρα να εισαγάγουμε έτσι αμερικανικά συστήματα κατά το οποίο δεν ισχύει. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Η πρώτη οδηγία του 2000 δεν είχε το αποτέλεσμα στην ε, επιχειρηματική ζωή που ήθελε Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν. Οπότε έχουμε εδώ πέρα μια επεξεργασία η οποία καλύπτει και μερικές νέες πτυχές. Σε αυτό προστίθεται και το πρόβλημα της ρευστότητας. Υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας πιστεύω σε κάθε κράτος μέλος, όχι μόνο στη δική μου χώρα, τη Γερμανία που το γνωρίζω, αλλά και σε κάθε χώρα κάποιες μικρές κυρίως επιχειρήσεις έχουν προβλήματα πέραν ε, από την οικονομική κρίση ε, και αυτό φτάνει μέχρι και την χρεοκοπία. Οπότε το αντιλαμβανόμαστε εμείς ε, εδώ πέρα και οι εισηγητές και θέλουμε πράγματι να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση αυτών ακριβώς των προβλημάτων της ε, ρευστότητα. Και επίσης μπήκαν εδώ πέρα και κάποιες διορθώσεις στη νέα αυτή πρόταση και νομίζω αναφέρεται σαφώς το έγγραφο εργασίας πως ε, η νέα αυτή οδηγία θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο μιας νέας κουλτούρας, αν θέλετε, της ε, δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης των ε, οικονομικών εταίρων. Αυτό από μόνο του βεβαίως δεν θα επαρκούσε, θα πρέπει να προσθεθούν και μια σειρά μέτρων πιθανώς από εθνική πλευρά και όχι μόνο από την ευρωπαϊκή πλευρά για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ανέφερα κάποια προβληματικά σημεία με την ε, πρόταση της ε, Κομισιόν. Ε, δεν συμφωνήσαμε οριστικά με τους σκιώδεις συγητές, όπως παραδείγματος χάρη η πρόταση της Κομισιόν να έχουμε υποχρεωτική ρύθμιση μόνο στις δημόσιες προμήθειες και στις ιδιωτικές συναλλαγές να έχουμε μια κάπως πιο ήπια υποχρέωση. Δεν πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό, πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να συμπεριληφθεί και ο ιδιωτικός τομέας, να έχουμε μια μορφή η οποία θα έχει μεγαλύτερο βαθμό καταναγκασμού από ό,τι προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Επίσης, ε, εκπληκτικό είναι πως ε, κατέδειξε η αξιολόγηση επιπτώσεων, πως υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν ε, καταγγέλουν ε, τους ε, ε, οφειλέτες τους γιατί και άρα δεν εμπεριέχονται σε αυτή την εικόνα εφόσον δεν έχουν καταθέσει κάποιες καταγγελίες. Οπότε προσπαθούμε εδώ πέρα να αντιμετωπίσουμε την όλη αυτή κατάσταση. Ε, ελπίζω και με τη βοήθεια του κλάδου και των αρμοδίων να γίνει αυτή μια εκστρατεία ενημέρωση έτσι ώστε και η μικρότερη επιχείρηση να γνωρίζει το τι μπορεί να ζητήσει και να απαιτήσει συμπεριλαμβανομένων και των τόκων σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση πληρωμής. Επίσης, αναφέρω μαζί με κάποιους άλλους ε, εισηγητές, εάν αφήσουμε εκτός τον ιδιωτικό τομέα, δεν έχει ακόμα καθοριστεί αυτό, αλλά δεν αποτελεί ε, και προτεραιότητα εδώ πέρα, πω ένα τμήμα ε, της οικονομίας, ειδικά αυτοί οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της ε, παροχής υπηρεσιών υγείας, σύνταξης κτλ. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν π.χ. όσον αφορά την σχετική ε, οδηγία περί προμηθειών, νομίζω 17 και 18 θα πρέπει... Στο 17 είναι, στο 18 θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Επίσης υπάρχει ειδική περίπτωση των νοσοκομείων σε κάποια, σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν ε, σε διάφορα νοσοκομεία, υπάρχουν διάφορα καθεστώτα, το ιδιωτικό και το κρατικό ή το περιφερειακό και υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των νοσοκομείων, δηλαδή τα νοσοκομεία αντιλαμβάνεστε πως έχουν μια ιδιαίτερη υποχρέωση παροχής ε, των υπηρεσιών, οπότε υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία και με τους σκιώδες συζητητές να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά τα νοσοκομεία εδώ πέρα. Τέλος, για το ύψος των αποζημιώσεων που προτείνει εδώ πέρα η Κομισιόν. και των πληρωμών και του λοιπού κόστους που έχει καταβληθεί. Έχουμε ακούσει τα επιχειρήματα υπέρ και κατά για το 5% αυτό το καταποκοπήν το εάν αρκεί. Οι μικρές επιχειρήσει λένε ότι είναι το ελάχιστο και λένε οι δήμοι από την άλλη μεριά πως είναι το, το μέγιστο. Πρέπει όμως να βρούμε ένα συμβασμό εάν θέλουμε να ε, ισχύσει κάποτε αυτή η οδηγία, οπότε αναμένω εδώ πέρα να ακουστούν επιχειρήματα για να βρούμε μία μέση οδό για να ισχύσει τελικά αυτή η οδηγία, γιατί είναι κάτι που απαιτείται άμεσα και δεν πρόκειται για κάποια έτσι ιδέα αφηρημένη της Κομισιόν είναι αποτέλεσμα του Small Business Act, είναι κάτι στο οποίο συνεισέφεραν πάρα πολλοί επιχειρήσει, είναι κάτι που ζήτησαν οι επιχειρήσει, δηλαδή να ισχύσει αυτή η οδηγία, να εφαρμοστεί ε, ένα σχετικό νομοθέτημα. Οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου όταν συζητάμε τις νομικές λεπτομέρειες. Σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν πάρα πολλές μικρές, μεσές και κάπως μεγαλύτερες επιχειρήσεις που ε, κινδυνεύουν και υποφέρουν από την καθυστέρηση πληρωμών των ε, εμπορικών τους ε, εταίρων και πρέπει και εμείς να κάνουμε ένα βήμα για να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Πάρα πολύ ξεκάθαρα μας τα είπατε και πολύ αξιόλογο το έγγραφο. Να δώσουμε τώρα την ευκαιρία στον κύριο Μπαλτασάρη να μας πει από πλευράς νομικής επιτροπής πώς έχουν τα πράγματα και κατόπιν έχουμε τους εμπειρογνώμονες. Κύριε Μπαλτασάρη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαιρετίζω την εκπρόσωπη της Επιτροπής, την κυρία Βάιλερ και τους συναδέλφους. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή διότι οργάνωσε την σημερινή συνάντηση. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε σε μια νομοθετική πρόταση που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κυρίως μια που μιλούμε για περίοδο ύφεσης και κρίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρόταση και δεν θα επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε η συντάκτης. Όμως, για να κάτσουμε και να επισημάνουμε μερικά σημεία πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε βέβαια τους ενδιαφερόμενους, έχουμε τους εμπειρογνώμας και έτσι ελπίζουμε να γίνει ένας διάλογος επικοδομητικός, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να υπάρξει μια ισόρροπη λύση όπως ακριβώς χρειάζεται. Πιο σημαντικές τώρα θα είναι οι κυρώσεις όσον αφορά την διοίκηση. Και η λέγει είναι ότι δεν υπάρχει η ίδια δυσκολία ε, οικονομική στη δίκηση όπως στις επιχειρήσεις. Και επίση υπάρχει, υπάρχουν πολλοί τρόποι χρηματοδότησης και εξεύρεσης πόρων από την διοίκηση. Και μιλούμε για ε, περίπου δύο δις που είναι τα, ο τζίρος της ε, συνεισφοράς της διοίκησης από το 2006 και μετά όσον αφορά όλη την Ευρώπη. Προβλέπεται εδώ μια προθεσμία 30 ημερών και κάποια άλλα μέσα, ούτως ώστε να μην έχουμε ε, πλέον άλλη τέτοια υπερημερία, τέτοια καθυστέρηση πληρωμών. Πάντως επιδίνονται κάποιες ε, δυνατότητες, κάποια περιθώρια παρεκκλήσεων. Θα πρέπει όλα αυτά να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα, ώστε να μην έχουμε κάποιο είδους λεόντιες ρήτρες. Συγκεκριμένα, κατά νου, έχω την δυνατότητα του σημείου 5 παράγραφος 3 σύμφωνα με την οποία διάταξη μπορεί να υπάρξει παρέκκληση αυτής της προθεσμίας των 30 ημερών εάν άλλος ορίζει η σύμβαση. Στο δε άρθρο 5 παράγραφος 4 είναι δυνατόν να έχουμε άλλες παρεκκλήσεις σε κάποιες ε, συγκεκριμένες συνθήκες. Εάν όμως όλα αυτά δεν διατυπωθούν με συγκεκριμένο τρόπο, τότε οι περίοδοι προθεσμίας των πληρωμών θα γίνουν ακόμα πιο μεγάλες. Βεβαίως, έχουμε την ελευθερία των συμβάσεων που είναι μια πάρα πολύ βασική αρχή του δικαίου. Θα πρέπει όμως αυτή η αρχή να περιχαρακωθεί με μεγάλη προσοχή. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος του να παρακάμπτει κανείς πάρα πολύ εύκολα την οδηγία. Επίσης θα πρέπει να υπόψη την κυρίαρχη θέση, τη δεσπόζουσα θέση της ε, δημόσιας αρχής, της διοίκησης, γιατί αποτελούν κάτι σαν ε, μονοπόλιο σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα ή τις ε, μικρότερες επιχειρήσεις. Τώρα, όσον αφορά κάποιες ασύμετρες, άνησες ε, διατάξεις ή όρους συμβάσεων, ε, αναφέρονται αυτό στο άρθρο 6. Επ' αυτού, νομίζουμε ότι θα πρέπει τα μέτρα τα προτινόμενα να αφορούν μόνο εξαιρετικέ περιπτώσεις που θα πρέπει και αυτές να οριστούν με σαφήνεια. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να οριστούν τα κριτήρια. Τα κριτήρια δυνάμει των οποίων μία τέτοια ρήτρα εάν επιβληθεί σε κάποιο συμβαλόμενο μέρος να θεωρηθεί ότι είναι άδικη και ετεροβαρής. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί το θέμα του κόστους της ίσπραξης θα πρέπει εδώ πέρα να δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται με το άρθρο τη πρόταση, γιατί έχουμε εδώ πέρα την παράγραφο 2, όπου λέει το πώ ορίζεται η δίκη και λέει ότι είναι κάθε είδου διοικητική αρχή ε, που ε, ε, περιγράφεται στην οδηγία του 2004 2018 Το πεδίο εφαρμογής, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2017 και συγκεκριμένα στο άρθρο 2. Σας ευχαριστώ. Well, thank you very much indeed, uh, I think for, uh, for, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες ε, παρατηρήσεις σας στους τομείς που αναφέρατε. Τώρα να αναφέρω το πρόγραμμα για το υπόλοιπο του πρωινού. Έχουμε τρεις ε, ειδικού θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Ο ειδικό από την Πολωνία δεν ήρθε να μιλήσει συγκεκριμένα για τον αντίκτυπο τις οδηγίες τους βασικούς ε, αποδέκτες της, ε, της μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οπότε θα δώσω τώρα στον λόγο στον κύριο Διάντζελη στο τέλος, γιατί ξέρω πως η Επιτροπή Μηχανίας ασχολείται ιδιαίτερα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν τους ειδικούς, μετά τον κύριο Διάντζελη και μετά τους συναδέλφους. Μετά το δεύτερο μέρος θα ακούσουμε εκεί εκπροσώπους ε, δημοσίων αρχών που ακούσατε ήδη από την εισηγήτρια πώς επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτές τις νέες προτάσεις και θέλουμε να τις ακούσουμε. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει η ακρόαση. Λοιπόν, από τους εμπειρογνώμονες έχουμε τον κύριο Μπεν Μπάτερς, Διευθυντή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ένωσης Επιμελητηρίων, Εμπορικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης. Έχουμε τον κύριο Χέντριξ, Διευθυντή Επιχειρηματικής Πολιτικής της ΟΕΑΠΜΕ που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες και μεταποιητικές επιχειρήσεις τον κύριο Ματέο Κάρλο Μπορσάνη από την Business Europe, Ένωση Επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ευρώπη. Ο καθένα σας λοιπόν έχει πέντε λεπτά και θα χρησιμοποιήσουμε και το χρονόμετρο για να το βλέπετε. Νομίζω εδώ πέρα η γραμματεία θα το χειριστεί. Ο καθένα λοιπόν έχει πέντε λεπτά χρόνο ομιλία και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Ντεάντζελη και τις υπόλοιπε ερωτήσει πριν περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Ο Μπεν νομίζω λοιπόν θα ξεκινήσει και θα... Μέχρι να βρούμε το δευτερόλεπτα, ε, μπορεί να, μπορεί να βρούμε το χρονόμετρο. Με συγχωρείτε, μπορεί να κερδίσει και κάποια δευτερόλεπτα. Very much. Malcolm, thank you very much. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρόσκληση και ευχαριστώ την εισηγήτρια ιδιαίτερα που μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ πέρα. Να συγχαρώ και την Επιτροπή για το πώς ε, χειρίζεται αυτόν τον φάκελο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ότι ξεκινήσατε αυτή την συζήτηση για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις κάτι το οποίο βεβαίως αποτελεί και πολύ καλό προηγούμενο για την Επιτροπή αυτή και για το Κοινοβούλιο συνολικά και είναι κάτι που πρέπει να επαναληφθεί. κυρία Βάιλερ ήδη έκανε κάποια σχόλια για το επίγον του πράγματος και θα ήθελα να το επαναλάβω και εγώ με το να σας δώσω κάποια στοιχεία από το δίκτυο μας. Εμείς κάναμε μία έρευνα την ε, Άνοιξη, την οποία επαναλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή και Μάρτιο-Απρίλιο τότε είχαμε πει πως ε, οι καστηριμένες πληρωμές από το δημόσιο τομέα είχαν αυξηθεί κατά 43% σχέση με τους προηγούμενους μήνες και ακόμη χειρότερα από ιδιώτες πελάτες είχε αυξηθεί η περίοδος πληρωμής κατά 60% σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Επίσης, ε, μας προξένει σε ιδιαίτερη έκπληξη το τι συνέβη με το δημόσιο τομέα, καθώς ε, φαίνεται πως είναι τελείως αντίθετο με τη φιλοσοφία προγραμμάτων ε, ανάκαμψης οικονομίας και τα μακροοικονομικά μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για να διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα δεν πληρώνουν εγκαίρως και πληρώνουν ακόμη πιο καθυστερημένα από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό είναι λοιπόν ανησυχητικό και πράγματι έχει δίκιο η συγγήτρια πρέπει να αναλυφθεί κάποια δράση και ταυτόχρονα δυσκολότερη γίνεται και η πρόσβαση στην πίστοση ε, ζητούνται με περισσότερες εγγυήσεις και κάποιες τράπεζες πολύ απλά δεν δίνουν τόσα δάνεια όσα έδιναν στο παρελθόν γιατί βεβαίω υπάρχουν και προβλήματα από την κατάρρευση των χρηματαγορών οπότε οι μικρομισές επιχειρήσεις πιέζονται και από τις δύο πλευρές. Οπότε εμείς θεωρούμε πως απαιτείται άμεση δράση εδώ πέρα και θεωρούμε πως η Κομισιόν καθυστέρησαν, η Κομισιόν καθυστέρησε στον συντάξει την έκθεση και βεβαίως μετά την ορμή που είχε δημιουργηθεί θέλετε από το Small Business Act καθυστέρησε πάρα πολύ η αναδιατύπωση. Κάτι το οποίο βεβαίω μετά έπεσε και πάνω στι ευρωεκλογέ, οπότε και το Κοινοβούλιο μπορούσε να κινηθεί μόνο μετά το καλοκαίρι, οπότε μείναμε πίσω γύρω στους 6 μήνες, κάτι το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, γιατί ήταν και στην κορύφωση της κρίσης. Οπότε πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για το εύρο τη οδηγία. Ε, θεωρούν πω καλύτερο είναι να μην το κάνουμε, γιατί αν αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα θα καθυστερήσουμε ακόμη περισσότερο και ίσως θα χρειαστεί να ξαναρχίσουμε την σύνταξη. Οπότε εμεί θα επικεντρωθούμε στην πρόταση τη Κομισιόν, την οποία καλωσορίζουμε, αλλά θεωρούμε πώ μπορεί να βελτιωθεί και όπω σα είπα, καλύτερο είναι να μην μπούμε στο ζήτημα τώρα του εύρου ε, τη οδηγία. αυτό θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Όπω είπα, καλωσορίζουμε την πρόταση της Κομισιόν. Η σχετική οδηγία είναι αναποτελεσματική, οπότε ήταν ε, απαραίτητη αυτή η αλλαγή. Θα κάνω τρία συγκεκριμένα σχόλια για το σχόλιο. Πρώτα απ' όλα για το περιεχόμενο, με συγχωρείτε. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζουμε τα βασικά στοιχεία τη ε, πρόταση που επικεντρώνεται στο ζήτημα των καθυστερημένων πληρωμών στι συναλλαγέ μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών. Καλωσορίζουμε την προθεσμία των 30 ημερών και οπωσδήποτε καλωσορίζουμε τη συμπερίληψη και των δημοσίων αρχών εδώ πέρα στην οδηγία. Ο κύριος Μπαλτασάρη αναφέρθηκε στις εξαιρέσεις για τις δημόσιες αρχές. Αυτό για μας είναι ζήτημα. Δεν θα λέγαμε, όπως ο κύριο Μπαλτασάρη πως δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία εξαίρεση στην προθεσμία των 30 ημερών και φαντάζομαι πως θα μας πούνε εδώ πέρα εκπρόσωποι των δημοσίων αρχών τα επιχειρήματά τους, δεν θα τα πω εγώ, αλλά θεωρούμε πως πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για το τι σημαίνει ε, το αιτιολογημένη εδώ πέρα όταν λένε πως μπορεί να υπάρχει μια αιτιολογημένη καθυστέρηση. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Γιατί όπως λέμε και στα αγγλικά δώσε θάρρος στο χωριάτι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, και βεβαίως πολύ περισσότερο όταν έχουμε εδώ πέρα αυτή την πολύ γενικόλογη έκφραση Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα πραγματικά να ξεκαθαρίσουμε το τι εννοούμε. Βλέπω πως έφτασα ήδη τα 5 λεπτά. Τελευταίο λοιπόν σημείο, αποζημίωση για το κόστος ανάκτησης. Το καταποκοπήν ποσό εδώ πέρα φαίνεται πως είναι δυσανάλογο. Πρέπει να υπάρχει ένα καταποκοπήν ποσό, αλλά πρέπει να είναι αναλογικό και με μια κλίμακα να αναλογεί προς το χρέος. Δεν μπορεί να έχουμε ένα, μια λύση για όλους. Και τέλος, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, θα θέλαμε τα κράτη-μέλη να λάβουν τα δικά τους μέτρα βράχη πρόθεσμα και ρεαλιστικά για να διευκολυνθεί η κατάσταση. Εμείς ως επιμελητήρια και οι λοιπές εμπορικές ενώσεις πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τις επιχειρήσεις. Να φέρω ένα ακραίο παράδειγμα. Εάν μια φιλανδική επιχείρηση πουλάει σε Έλληνα πελάτη πρέπει να γνωρίζει πως η περίοδος πληρωμής διαφέρει πάρα πολύ από αυτή που έχουν συνηθίσει όταν κινούνται εντός φιλανδικής αγοράς. Πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε κι εμείς για να αποφύγουμε αυτές τις ανησυχητικές τάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λέει και ο Πρόεδρος και ευχαριστώ που τηρήσατε και το, τον χρόνο για τις παρατηρήσεις σας προς τα κράτη-μέλη και εγώ θα ήθελα να βρίσκεται εδώ πέρα το Συμβούλιο βρίσκεται η Σουηδική Προεδρία και είμαι σίγουρος ότι σας ακούει και η Ισπανική οπωσδήποτε θα σας παρακολουθεί πολύ στενά. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον κύριο Λουκ Χέντριξ να περάσουμε παρακάτω. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να συγχαρώ και εγώ τον ε, εισηγητή για την πρωτοβουλία αυτής της, μήνυ, της διοργάνωσης αυτής της ακρόασης και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Όπως είπε και ο εισηγητής, οι καθυστερήσεις πληρωμών μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο με έναν ευρύ φάσμα συμπληρωματικών μέτρων. Όλοι συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων επιχειρήσεων και των ίδιων των επιχειρήσεων πρέπει να αναλάβουν ευθύνε. Ιδάλω, η νομοθεσία μόνο της δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Το νομικό πλαίσιο οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθεί σε κάθε περίπτωση. Παρά τις καλές προθέσεις και τις αξιέπαινες προσπάθειες της Επιτροπής, η πρόταση δεν είναι ιδανική για τις μικρές επιχειρήσεις. Απέχει πολύ από αυτό. Γι' αυτό έχουμε τέσσερις σοβαρές παρατηρήσεις και απαιτήσει σχέση με την πρόταση. Πρώτα απ' όλα για το πεδίο, το, την, ε, το κομμάτι επιχειρήσεις προς πελάτη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων προστατεύονται ε, όλες ανεξαρτήτως, χωρίς εφόσον πρέπει να πληρωθεί ένα τιμολόγιο και εφόσον εμπλέκεται ένας καταναλωτής. Η κοινή πρακτική μεταξύ καταναλωτών είναι να μην καταβάλουν το σύνολο του ποσού και να περιμένουν να δρανήσει η επιχείρηση. Συνήθως δεν υπάρχει προσφυγή. Οι καθυστερήσεις λοιπόν πληρωμής ε, στο B2C ε, αφορούν ιδιαίτερα τον ε, τομέα των μικρών επιχειρήσεων και τον κατασκευαστικό τομέα. Σε αυτήν την περίοδο κρίσης πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να αποφύγουμε τέτοιου είδους δυσκολίες. Θα πρέπει να έχουν όλοι το απαραίτητο μετρητό για να πληρώσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους. Ε, εδώ πέρα δεν έχουμε λάβει παρκώ υπόψη την προστασία των καταναλωτών όμω στην πρόταση τη οδηγία. Διότι οι καταναλωτέ έχουν και θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και θεμελιώδει υποχρεώσει. Τώρα μια παρατήρηση για τον δημόσιο τομέα. Ο κ. Μπαλντασάρη ήδη το σχολίασε. Σε περίοδο κρίση πρέπει κανεί να αγωνιστεί για να κρατήσει την απασχόληση σταθερή. Είναι απαράδεκτο λοιπόν οι δημόσιε αρχέ να έχουν καθυστερήσει στι πληρωμέ. Ε, εκτιμούμε τι ε, προσπάθειες της Επιτροπής να μειώσουν τις προθεσμίες πληρωμής για τις δημόσιες αρχές, όμως αυτό δεν αρκεί καθώς δεν υπάρχει μέγιστο όριο. Ιδίω ε, για την υπέρβαση των 30 ημερών, το προτινόμενο κείμενο δεν απαγορεύει στα κρατημέλη να πληρώσουν μετά από 30 μέρες. Ε, αυτό είναι ακόμη επιλογή. Οι δημόσιες αρχές λοιπόν, οι κρατικέ αρχέ θα πρέπει να παρατείνουν τους όρους πληρωμής όταν μπορούν να αιτιολογήσουν αντικειμενικά την απόφασή τους Και μεταξύ των μερών θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ελευθερία ώστε να μην ε, επιτρέπονται τέτοιου είδου στρεβλώσεις των πληρωμών. Θα πρέπει να ε, δούμε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσει διαπραγματευτικές δυνάμεις ε, των κρατικών αρχών τέτοιε που καθιστούν την ε, ελευθερία των συνελλαγών μια πραγματική φαντασίωση. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι οι υποχρεώσει που επιβάλλονται στι κρατικέ αρχέ είναι πολύ ασαφεί και θα παραβιαστούν από τι δημόσιε αρχέ. Πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη αιτιολόγηση για να είναι υπόλογε με τον ίδιο τρόπο όπω όλοι οι υπόλοιποι και οι κρατικέ αρχέ. Επί τη αρχή λοιπόν θέλουμε μια ε, συγκεκριμένη περίοδο 30 ημερών και αν πρέπει να δεχτούμε εξαίρεση, ίσως κάποιο να έχει περισσότερη φαντασία από μένα, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει λόγο να δεχτούμε εξαιρέσει. Αν αυτέ πρέπει να υπάρχουν, τότε να δικαιολογούνται αναλόγω και σε κάθε περίπτωση να περιορίζονται στις 60 ημέρες. Η τρίτη μου παρατήρηση, οι σχέσεις B2B, επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις, τα δικαιώματα αντιστάθμισης για το κόστος ανάκτησης και ε, το να επιτραπεί στους ε, πιστωτές να καθυστερήσουν τις πληρωμές είναι κάτι που καλωσορίζουμε. Όμως θα πρέπει να προβλεφθεί και μια σχετική υποχρέωση. Θα πρέπει να υπάρξει επιβολή τόκου σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών και αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό για τις μικρές επιχειρήσεις δεδομένων των εμπορικών του σχέσεων με τις μεγαλύτερες ε, επιχειρήσεις. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η περίοδος εντός της οποίας οι επιχειρήσεις πληρώνουν τις άλλες επιχειρήσεις και αυτή η περίοδος θα πρέπει μέσα στην οδηγία να περιορίζεται σε ένα μέγιστο όριο των 60 ημερών. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο, διότι η οδηγία δεν απαγορεύει την παραβίαση ελευθερίας ε, συναλλαγματικής των πιστωτών. Αυτό έχει επιδεινωθεί λόγω των συνδικών της κρίσης. Οπότε βλέπουμε ότι οι, μικροεπιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προχρηματοδοτούν κάποιες δραστηριότητε τους. Σήμερα δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει ελευθερία στις συναλλαγές, διότι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τόσο μεγάλη δύναμη που οι μικρομεσαίες δεν έχουν καμία δυνατότητα διαπραγματευτική πλέον. Πολλέ φορέ χρησιμοποιείται το επιχείρημα ότι αυτό θα έχει συνέπειε και για άλλα διαπραγματευτικά σημεία μεταξύ επιχειρήσεων, όπω οι τιμέ, η εκτόσεις, αλλά αυτό δεν ε, είναι βάσιμο σε επιχείρημα. Διότι ως σήμερα οι μεγάλες επιχειρήσεις παραβιάζουν και εκμεταλλεύονται τη θέση τους προκειμένου να πιέσουν ως προμηθευτές. Έπειτα η μείωση του μέγιστου ορίου πληρωμής ε, στις σχεσεις b B2B θα πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστεί. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ σαφή και συνολική παρουσίαση. Τελευταίος μας ομιλητής, αυτό το τμήμα της ακρόασης, ο κύριος Μποζάνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ετοιμάσει μια παρουσίαση PowerPoint, πολύ σύντομη. Θα σας διατεθεί. Με... Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω το ζήτημα αυτό, αυτή τη σοβαρότατη πρόταση. Το όνομά μου είναι Ματέο Μπορσάνη, εργάζομαι για την Κονφιντούστρια στις Βρυξέλλες. Είμαστε το μέλος από την Ιταλία της Business Europe. Γιατί μιλάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα. Μιλάμε για ένα σημαντικό ποσό οικονομικό. 180 δις ευρώ θα διατεθούν στις επιχειρήσεις εάν οι δημόσιες αρχές πληρώσουν τους εκκρεμείς λογαριασμούς τους μέσα σε 30 ημέρες. Αυτό ορίζει η πρόταση. Στην Ιταλία και μόνο, εάν τη δούμε ως παράδειγμα, 60 δις ευρώ πιστώσεων των εταιριών ω προ τι δημόσιε αρχέ οφείλονται ακόμη και 5, 40 μάλλον δι αφορούν μόνο τον τομέα τη υγεία, τον πιο κρίσιμο. Για να κάνουμε μια άμεση σύγκριση, 5 δι ευρώ, 12 φορέ λιγότερα, είναι το ποσό που η Ιταλική κυβέρνηση παρέχει και προβλέπει για να ανακάμψει από την κρίση. Πολύ σύντομα στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τις μέσες πληρωμές σε 30 ημέρες από τις δημόσιες αρχές προς τις επιχειρήσεις. Θα δείτε και στην επόμενη διαφάνεια ότι στην πραγματικότητα έχουμε τρία κράτη-μέλη τα οποία ήδη ακολουθούν λίγο πολύ τις προδιαγραφές της πρότασης. Όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να βελτιώσουν πολύ σημαντικά την συμπεριφορά τους ως προς τις πληρωμές, ιδίως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιταλία. Εάν δείτε τον τομέα της υγείας, που όπως είπα είναι ο πιο κρίσιμος, θα το δείτε και στην ερχόμενη διαφάνεια, οι αριθμοί είναι πολύ πιο ανησυχητικοί. Το 2009 έχουμε ένα μέσο όρο 300 ημερών καθυστέρησης. Και παρόλα αυτά, αυτά είναι τα εθνικά μόνο δεδομένα. Αν δεν κανεί τα περιφερειακά, δεν τα συμπεριέλαβα γιατί είχα μόνο 5 λεπτά, οι καθυστερήσει φτάνουν τι 600 ημέρε. Εάν λοιπόν όλα αυτά ληφθούν υπόψη ταυτόχρονα, το πρώτο μας σχόλιο είναι ότι γενικώ στηρίζουμε την πρόταση και γενικώ πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ των σχέσεων B2B και B2 Public Authorities, ε, ε συμβάσεις αυτές. Γιατί θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Οι δημόσιες αρχές δεν μπορούν να δεσμευτούν σε μια σύμβαση χωρίς να έχουν προπολογισμό και εξάντε ποσά. Έπειτα, διότι οι δημόσιες αρχές έχουν ροή πρέπει να έχουν μια σταθερή ροή εισοδήματο και την έχουν χάρη στου φόρου. Και έπειτα γιατί οι, πληρωμέ, οι καθυστερήσει πληρωμών είναι πολύ μακρύτερε. Άρα, εάν η ασθένεια είναι σοβαρότερη, ακόμη και το φάρμακο θα πρέπει να είναι πιο δραστικό. Δεύτερο σχόλιο δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων εταιριών. Αυτό θα ήταν σφάλμα, διότι θα προκαλούσαμε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι μικρομεσαίε είναι σταθεροί προμηθευτέ των μεγάλων εταιριών στι ε, ολοκληρωμένε αλυσίδε παραγωγή και υπάρχουν τέτοιε συμβάσει και προμήθειε που θα ήταν ανέφικτο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει να συμμορφωθούν με τέτοιε υποχρεώσει. Εφόσον ε, συνεργάζονται με μεγάλε εταιρείε, πώ θα τα έβγαζαν πέρα. Ένα άλλο σχόλιο το είπε και ο προηγούμενος ομιλητής και συμμερίζομαι πολύ το έργο του και τα σχόλιά του. Δεν θα πρέπει να προβλέψουμε καμία εξαίρεση για συγκεκριμένους τομείς. Εδώ θα ανοίγαμε ένα κουτί της Πανδώρας και αν τα ανοίξουμε θα αποδυναμώσουμε την ουσία της πρότασης. Αντιθέτως, θα έπρεπε να βελτιώσουμε τη διατύπωση και την δομή του άρθρου 5. Και ως προς το κείμενο, διότι πρέπει να αποσαφινιστεί και ως προς την διάρθρωσή του. Εάν, και το τονίζω, εάν δικαιολογείται να έχουμε μακρύτερες περιόδους, αυτό θα πρέπει να δικαιολογείται βάσει της αρχής της αναγκαιότητας, κάτι που μου φαίνεται από νομικής άποψης περισσότερο δεσμευτικό. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να παραβαίνουμε τα σταθερά όρια. Και μια τελευταία παρατήρηση χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση. 30 ημέρε, ναι, αλλά ημερολογιακέ ή εργασίε. Εγώ φαντάζομαι ότι η πρόταση τη Επιτροπή εννοεί ημερολογιακέ, ε, αλλά ίσω και ήταν καλύτερα να διευκρινιστεί. Επίση, ο ορισμό των δημόσιων αρχών. Ε, και αναφέρονται αυτέ και στο άρθρο 1,9 του κανονισμού 18 και στο άρθρο 2.1 της Οδηγίας 17 για τις δημόσιες προμήθειες. Ίσως να ακολουθήσουμε αυτούς τους ορισμούς. Επίσης να βελτιώσουμε τη διάρθρωση των άρθρων, ιδίω το 3 και 4, τα οποία αναφέρονται μόνο στις συμβάσεις μεταξύ εκμεταλλεύσεων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπορσάνη. Όχι μόνο μιλήσατε ακριβώς πέντε λεπτά, αλλά μας προτείνατε και καταπληκτικές λύσεις. Ελπίζουμε ότι οι 250 ημέρες στο μέσο όρο πληρωμής των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ιταλία θα διορθωθεί. Ίσως ο κύριος Καρέλ να έχει κάποια σχόλια στη συνέχεια. Τώρα θα ανοίξουμε τη συζήτηση και θα ακούσουμε ερωτήσεις. Ο κύριος Ντεάντζελης θα ήταν καλό να μιλήσει για την διάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ίσως τον αφορά ιδιαίτερα στο ζήτημα αυτό. Και έπειτα θέλω να δω κατά πόσον οι συγκητές θέλουν να παρέμβουν. Έχω τον κύριο Κόρτσμαν. Θέλετε να θέσετε ερώτηση. Η κυρία Ρούλα, ο κύριος κοζίφνικ Έχουμε και άλλους ομιλητές από την Επιτροπή μας. Τον κύριο Γκέπχαρτ, Σβάρπ, Μπεζόη. Έχουμε πολλούς ε, παρεμβαίνοντες. Θα ζητήσω λοιπόν να είστε αρκετά σύντομοι στις ερωτήσεις σας για να προλάβουν οι ομιλητές να απαντήσουν. Κύριε Ντεάντζελης, θέλετε να ξεκινήσετε ως εισηγητής ε, εκ μέρους της Επιτροπής Βιομηχανίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω την κυρία Βάιλερ, την εισηγήτρια για τις προσπαθίες της και ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον πρόεδρο που μας προσέφερε αυτήν την ε, διοργάνωση της ακρόασης, της συζήτησης για ένα θέμα τόσο πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Σήμερα το λεγόμενο ρίσκο της επιχείρησης, ο κίνδυνος επιχείρησης στην Ευρώπη παρουσιάζει παράγοντες και στοιχεία που κάποιες φορές είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ κρατών. Κάποια παραδείγματα ήδη αναφέρθηκαν, διότι κάποιος που έχει μια επιχείρηση στη Δανία και πρέπει να λάβει πληρωμές ε, για τις πρώτες ε, μέσα σε 36 μέρες πρέπει να σεβαστεί αυτό το λογαριασμό ενώ οι ίδιες προϋποθέσεις σε, άλλε, σε άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία ή την Ελλάδα σημαίνουν ότι θα πρέπει να περιμένει ο ίδιος άνθρωπος 155 ημέρες. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα στην Ιταλία. Μας, ε, μας υπενθυμίστηκε η κατάσταση του τομέα της υγείας που είναι δύσκολη και ευαίσθητη. Έχουμε ένα μέσο όρο 138 ημερών ενώ έχουμε 68 ημέρες μέσω όρο στην Ευρώπη. Κατά τα άλλα, ενώ έχουμε μέσους όρους στην Ισπανία και την Ελλάδα μεγαλύτερους, αυτό δεν σημαίνει ότι το ζήτημα δεν πρέπει να επιληθεί. Γιατί τώρα αυτή η μελέτη του θέματος, γιατί υπάρχει τέτοια ανομοιότητα στο πώς γίνονται οι πληρωμές. Κατά την άποψή μας, Υπάρχει ένας, αυτό είναι ένας παράγοντας ανασταλτικός για την εσωτερική μας αγορά. Η έλλειψη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων χωρών επιβάλλει στον Ευρωπαίο νομοθέτη να αναλάβει δράση για αυτό το περίπλοκο ζήτημα των ε, κανόνων για τις εθνικές συμβατικές υποχρεώσεις. Θα ήθελα να σταθώ στην πτυχή που θεωρώ πολύ σημαντική περισσότερο από κάθε άλλη μάλιστα, και που απειλεί το μέλλον των επιχειρήσεών μας. Λόγου χάρη, η δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις δραματική έλλειψη ρευστού μετρητών. Αυτό επιβάλλει έναν αριθμό και δυσκολεύει έναν αριθμό αυξανόμενο και πολύ σημαντικό μικρών, ε, μεσαίων και ιδιαίτερα μικρών επιχειρήσεων της Ευρώπης. Είναι θέμα σοβαρό, όπως και η πρόσβαση ε, στις πιστώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η οικονομική κρίση και η συρρήκνωση οικονομική των τελευταίων μηνών είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί εδώ καθορίζουμε το μέλλον του παραγωγικού και βιομηχανικού και επιχειρησιακού μας κόσμου στην Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι για, να... για μια μικρομεσαία επιχειρήση είναι πολύ δύσκολο και κοπιαστικό να φτάσει στις τραπεζές μαζικές ε, πιστώσεις και να έχει πρόσβαση σε αυτές και με όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις που τη βαρύνουν και τους λογαριασμούς ε, τελικά καταλήγει να γίνεται πληρωμή με πάρα πολλούς μήνες καθυστέρησης. Αυτή λοιπόν, ε, αυτός είναι ο λόγος που ω εισηγητή τη Επιτροπή τη Βιομηχανία δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω την πρόταση τη Επιτροπή. Θεωρώ ωστόσο ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Η οδηγία 35 του 2000 είχε αντίκτυπο ε, πολύ μέτριο. Θα πρέπει λοιπόν η νέα οδηγία να είναι αποτελεσματική και επιτυχής και να, να περιλάβει στοιχεία σαφήνειας και ορθότητα και διόρθωση των εμπορικών σχέσεων και των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αγωγής, της ε, αναθεώρησης των ορών πληρωμής και του υπολόγου των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να δούμε την ανάγκη ώστε να φτάσει ως μέγιστο όριο η προθεσμία των 30 ημερών. Θεωρώ ότι η θέση σε ισχύ των ε, υποχρεώσεων που προβλέπει η οδηγία είναι σημαντική για το έγκαιρο των ε, πληρωμών. Άλλωστε, οι προτάσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ένωση τους στην Ευρώπη έχουν κάνει ανάλογες προτάσεις και θέλουμε να καλυφθούν εδώ όχι μόνο οι σχέσεις μεταξύ δημόσιων αρχών και επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων και επιχειρήσεων, αλλά και επιχειρήσεων με καταναλωτές. Είναι σημαντικό αυτό γιατί είναι πρωτογενή πηγή εσόδων για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει τη Ευρώπη. Σε σχέση λοιπόν με την πρόταση αυτή, νομίζω ότι το θέμα θα πρέπει να το δούμε χωρίς να παραβλέπουμε και την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Άρα η επιλογή της Επιτροπής να, προτα... να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης είναι μια πρόταση που συμμεριζόμαστε. Όμως το νομοθέτημα, το κοινοτικό θα πρέπει να συμβάλλει έτσι ώστε να έχουμε βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου γενικότερα. Οι κανόνες και οι εξαιρέσεις για τους όρους πληρωμών θα είναι ένα σημείο το οποίο θα καθορίσει το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Κύριε Ντιάντζης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τις προτάσεις σας, τις προτάσεις της Επιτροπής της Βιομηχανίας. Και τώρα να προλάβουν το λόγο οι σκιώδεις ηγετές. Ε, αυτοί έχουν την προτεραιότητα, αλλά να δούμε ποιοι άλλοι μπορούν στη συνέχεια να μιλήσουν. Ε, αν υπάρχει κάποιο είδους ερώτηση. Ο σκιώδης ηγετής του ΕΛΚ πρώτος ίσκυοδης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει η κυρία Χάντσλικ. Ευχαριστώ και όσους ε, μας μίλησαν και μας ενημέρωσαν σήμερα. Οπωσδήποτε αυτή η πρόταση είναι σημαντική όσον αφορά το τι θα γίνει με τις ΜΜΕ σε σχέση με τις δημόσιες αρχές. Έχω μία ερώτηση προς ε, τον κύριο Χέντες. Δεν κατάλαβα αν σας κατάλαβα καλά. Το περίφορο εφαρμογή της οδηγίας είναι δυνατόν να παρεκταθεί και για τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και για τις δημόσιες αρχές. Καλά κατάλαβα. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, θα καλύπτονται και αυτές οι συμβάσεις, δηλαδή η μεταξύ επιχειρήσεων. Και σε αυτή την περίπτωση, μήπως φοβάστε ότι η ελευθερία των συμβάσεων των ΜΜΕ πρόκειται να περιοριστεί. Άλλη μια ερώτηση από του υπόλοιπου Αυτές οι δαπάνες ανάκτησης δεν θα πρέπει να ρυθμιστούν με διαφοροποιημένο τρόπο σε σχέση με το κατά περίπτωση ποσό ή θα πρέπει να υπάρχει ένα ποσό συγκεκριμένο. Τι λέτε. Βάιλα, για πέστε μου, κυρία. Ε, είπατε να έχουμε ένα, ποσό, ένα ποσοστό φίξαν συντελεστή 5%. Ε, αν έχουμε όμως μια δημόσια σύμβαση ας πούμε του ύψου των 20 εκατομμύριων ευρώ τότε αυτό το 5% της εν λόγω σύμβασης είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Άρα μήπως αυτό το καταρχήν καταποκοπή ποσό θα πρέπει να αυξομοιωθεί ανάλογα με την περίπτωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Ελπίζω ότι η συζήτησή μας θα είναι όσο γίνεται πιο δημιουργική. Ο Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε. Πρέπει να αναφροντίσουμε να υπάρχει χρόνος να μιλήσουν όλοι, όλοι. Κύριε Κρότσμα, έχετε πρώτο το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Κρότσμαν. Με συγχωρείτε, ευχαριστώ πράγματι αναφέρθηκε το πώς θα πρέπει να επεκταθεί η οδηγία και στον καταναλωτή. Πώς θα γίνει οι καταναλωτές είτε μετρητά πληρώνουν είτε με πιστοτικές. Και αν δεν έχουν ε, εταιρεία, εντάξει, συνήθω, όταν ε, έχουν κάποιου χειρόνακτες που εργάζονται για αυτού, ε, συνήθω έχουν μια προθεσμία 30 ημερών. Δεύτερον, είπατε πώ πρέπει να επεκταθεί στι συναλλαγέ μεταξύ επιχειρήσεων μήπως είναι πιο λογικό αυτό το οποίο είχε προταθεί δηλαδή να πούμε πως ισχύει για τον δημόσιο τομέα όχι μεταξύ επιχειρήσεων αλλά να υπάρξει μία μέγιστη προθεσμία των 60 ημερών. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα των μικρών επιχειρήσεων ε, καθώς συχνά πληρώνουν, συναλλάσσονται με συγχωρείτε μεγάλες επιχειρήσεις και δεν μπορούν να διαπραγματευτούν τους όρους. Οπότε νομίζω θα τους βοηθούσε να βάλουμε εκεί μια μέγιστη προθεσμία 60 ημερών και εντός των 60 ημερών υπάρχει η ελευθερία του τι συμφωνία θα κλείσουν. Και τέλος για το κόστος αυτό που είπατε νομίζω πως θα έπρεπε να είναι κάπως κλιμακωτό γιατί βεβαίως το κόστος ε, το διαδικαστικό είναι ίδιο είτε μιλάμε για 10 ευρώ χρέος είτε για 10.000 ε, ευρώ χρέος. Οπότε πως θα ήταν σωστότερο να πούμε πως ε, το 40 ευρώ να είναι διοικητικό κόστος π.χ. για όλα τα, τα χρέη και να μην έχουμε ένα 5% ως ε, κύρωση και μετά να λέμε πως είναι μεγάλο το ποσοστό όταν μιλάμε για τα μεγάλα πως Εάν υπάρχει μετά κάποια παράβαση να υπάρχει μια δεύτερη, αν θέλετε, προσάρξη. Αυτές τις ερωτήσεις είχα ευχαριστώ. Uh, Κυρία Ρούλε. Πρώτα απ' όλα είπατε περί διεύρυνσης ε, του πεδίου. Θα έχουμε πάρα πολλές διαπραγματεύσεις και μεγάλη καθυστέρηση. Αν μειωθεί επίσης ε, το εύρος, έχουμε δει πως ε, στο παρελθόν η σχετική οδηγία νομίζω ήταν αρκετά περιορισμένη στην παλιά πρόταση. Στη νέα οδηγία έχει διαγραφεί και μια οδηγία περί ε, δημοσίων προμηθειών και αναρωτιέμαι γιατί συνέβη αυτό. Εγώ νόμιζα πως θα έπρεπε να υπάρχει ε, να παραμείνουμε σε αυτά τα οποία έχουμε. Δεν πρόκειται για κάποια διεύρυνση. Νομίζω μένουμε σε αυτά τα οποία ήδη καλύπτονταν και θα δημιουργούσαμε σοβαρότερο πρόβλημα με βάση τι εμπειρίες που έχουμε αν την περιορίζομαι. Κατά τα λοιπά συμφωνώ με τους ε, προλαλήσαντε και θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα του 5, ε, του 100 και ταυτόχρονα την κλιμάκωση. Δεν το βρίσκω, να σου πω την αλήθεια, αναλογικό με το πρόβλημα που υφίσατε και νομικά προβληματικό, να σα πω την ειλικρινή μου άποψη. Ευχαριστώ, κύριο Σκοτσίσνικ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω κάτι να ρωτήσω την κυρία Βάλε την συγκεντριά μας γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα δημιουργεί κάποιο πρόβλημα ε, ε, από αυτό το ζήτημα, το οποίο βέβαια η ίδια πάρα πολύ καλά το μελέτησα και εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να διερευνήσουμε τα τι ρωτήματα ανακύπτουν. Τώρα, η ερώτηση μου είναι εξή, μια που κάνω αυτή την ε, ε βέβαια να ευχαριστήσω και να συγχαρώ πρώτα πρώτα-πρώτα τους συζητητές Είναι θέμα καυτού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ποια είναι η ερώτηση. Η ερώτηση είναι η εξή. Η περιμερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετική σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους ιστορικούς, σε ορισμένες χώρες. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορούσε να αποδώσει και να λειτουργήσει έβδομα μια τέτοια ρύθμιση. Ευχαριστούμε, λέει ο Ακούσαμε τις ερωτήσεις όλων των ισχυωδών εισηγητών και τώρα, εάν συμφωνούν οι συνάδελφοι, θα ήθελα να δώσουμε την ευκαιρία στους τρεις μας συμπληρογνώμενες να μας δώσουν κάποιες σύντομες απαντήσεις όσο ρωτήθηκαν. Και κατόπιν να πάμε στο επόμενο τμήμα της ε, ακρόασης. Εντάξει, αν δεν έχετε αντίρρηση. Μην ξέρω αυτός αν κάποιος άλλος έχει ε, κάποια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη στους ε, ε, συζητητές. Α, πολύ ωραία. Πετε μας αν μπορείτε τι απαντήσει έχετε για όσα ερωτήθηκαν. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μπάντες, πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, όσο μας είπαν ε, οι βουλευτές και όσον αυτό το 5% και όσον την, την, την κύρωση και όχι εγώ λέω να μην έχουν χαρακτήρα κυρωτικό, χαρακτήρα κύρωσης και τιμωρίας θα πρέπει να είναι κάποιο είδους αντιστάθμιση, αποζημίωση τέτοιο χαρακτήρα να έχει και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα είναι φίξη ή όχι το επίπεδο ε, και τελικά να είναι αναλογικό. Δηλαδή, λόγω της περιμερίας να εξετάσουμε πόσο ζημιώθηκε ο πιστωτής. Επίσης, είπαμε αυτό το 5% ε, επιπλέον ίσως ε, αποτελεί μια παράδοξη, μια περίεργη ε, προσέγγιση και έτσι έχει προοδευτικό χαρακτήρα και όχι δεν, δεν είναι ένα καθορισμένο ποσό σταθερό. ο τελευταίος ε, ομιλητής μας είπε κατά πόσον ε, και αυτό το νομοθέτημα θα μπορέσει να αποδώσει όλες τις χώρες. Για την αλήθεια ότι έχουμε πολύ διαφορετικό τοπίο σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Άρα, αυτό είναι μια ολόκληρη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πάνω σε αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε. Κύριε Χέντριξ, υπήρχε κάποια ερώτηση ακριβώ σε εσά ε, συγκεκριμένα. Σα ευχαριστώ. Λέει ο κύριο Χέντριξ, ε, σε σχέση με τι συμβάσει επιχείρηση με επιχείρηση. Ναι, ναι, καλά καταλάβατε κυρία. Ήδη καλύπτονται αυτού του είδου οι συμβάσει από την οδηγία. Όμω αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να τεθεί ένα όριο χρονικό, μάξιμουμ όσον αφορά τέτοιου είδους ε, συμβάσεις. Αυτό ανατρέπει την ελευθερία των συμβάσεων. Όχι. Χρειάζεται όμω μια ρύθμιση που να μπορεί να καλύψει και τι ΜΜΕ, γιατί γνωρίζετε ότι εμεί από πλευρά του δικού μα φορέα πάντα θέλουμε να υπάρχει ελευθερία των συμβάσεων, αλλά θα πρέπει κάτι να γίνει τώρα, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία συμβάσεων όσον αφορά τι συμβατικέ σχέσει των επιχειρήσεων μεταξύ του. Τώρα, όσον αφορά αυτό το ποσό, το καταποκοπή, Έχουμε αυτά τα 40 ευρώ, αυτό αναφέρεται και στην έκθεση της κυρίας Βάιλερ. Ίσως σε κάποιες χώρες αυτό το ποσό δεν αργεί. Όμως υπάρχει ε, και η δυνατότητα να έχουμε επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στις δαπάνες ανάκτησης και να συζητηθεί τώρα κατά πόσο βέβαια αυτό θα πρέπει να είναι λογικό ή όχι. Πάντως σας τονίζω ότι όταν μιλούμε για επιπλέον κόστος ε, ανάκτησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι συνήθως οι νήμοι ε δεν αναθέτουν ε, κάποιες ε, ενέργειες σε εξωτερικές εταιρείες. Δεν κάνουν το outsourcing. Και το θέμα είναι κατά πόσον αυτό του, οι δαπάνε επιπλέον είναι εδώ να, να αποδειχθούν. Α πούμε, από ένα δικηγόρο αποδεικνύεται η δαπάνη, αλλά όχι πάντα. Τώρα, για το κατά πόσο θα πρέπει να βιαστούμε ή όχι. Ναι, ναι, βεβαίω και το θέμα αυτό επήγε. Και από την άλλη μεριά όμω προτιμούμε να είναι άρτια, επιτυχημένη η νομοθεσία. Να μην είναι κάτι το οποίο έγινε στο γόνατο. Γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι η οδηγία ήδη θα πρέπει να έχει γίνει και να έχει ε, αναθεωρηθεί εδώ και μια πενταετία. η δε νέα οδηγία θα υποστεί αναθεώρηση σε δύο χρόνια. Μπορζάνι, να στα πω στα ιταλικά. Σε ό,τι αφορά το κόστος ανάκτησης, συμφωνώ με όσα μόλις είπε ο κύριος Ένριξ. Τα 40 ευρώ είναι απλώς μια συμμεβαστική λύση, ένα σημείο ισορροπίας το οποίο μπορεί να μεταβληθεί ή και όχι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Για το 5% και εδώ, κατά την άποψή μου, το ποσοστό είναι αποδεκτό, είναι ισόρροπο. Αλλά δεν είναι και επιτακτική ανάγκη. Μπορεί να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Κατά την πορεία που θα ακολουθήσει η εξέταση πρόταση του Κοινοβουλίου. Το σημαντικό είναι να μην υπάρξουν αποκλεισμοί εξαιρέσει. Δεν θα πρέπει να υπάρξει τιμωρητική χρήση. Κανεί δεν θέλει να τιμωρήσει τα κατημέλη, ούτε τι επιχειρήσει, αλλά θα πρέπει να γίνονται συμβαστοί οι όροι των συμβάσεων. Αυτό ισχύει και για τι επιχειρήσει και για τα κράτη-μέλη. Εκεί που το πρόβλημα είναι οξύτερο για τα κράτη-μέλη θα πρέπει τα μέτρα να είναι πιο ασφαλή, πιο δεσμευτικά. Ιδάλω επιστρέφουμε στο σημείο αφετηρία του 2035, που τελικά δεν έφερε κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι τα είπα όλα προς στιγμή. Σας ευχαριστώ και τους ε, τρεις γιατί μας δώσατε χρήσιμες πληροφορίες. Θα ήθελα τώρα να περάσω στους επόμενους εμπειρογνώμονες. Απλά θα ήθελα να πω στους συναδέλφους πως έχω για τους επόμενους ομιλητές, κύριος Γκέπχαρτ Φαπόσελτ και Μπονιέ. Αν θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει στον κατάλογο, να μας το πει. Α, ο κ. Τζιούν ήρθε, ο σκιώδης εισηγητής. Έπρεπε να έχετε έρθει λίγο νωρίτερα βεβαίω. αλλά οπωσδήποτε θα μιλήσετε κι εσείς. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο επόμενο, στην επόμενη φάση των εμπειρογνωμόνων για το τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στις δημόσιες αρχές. Καλωσορίζω λοιπόν πρώτα απ' όλα τον κύριο Όλαφ Μόμπεργκ από τη Σουηδική Ένωση ΟΤΑ είχαμε την ευκαιρία να σας συναντήσουμε στην Σουηδία και χαιρόμαστε που σας καλωσορίζουμε και εδώ πέρα και γιατί βεβαίως Σουηδία αυτή τη στιγμή έχει την Προεδρία. Μετά είναι ο κύριος Γκίντ Πφούντστάιν ε, από την Γερμανική Δευτεροβάθμια Ένωση Δήμων. Ναι, με συγχωρείτε για την προφορά μου στα γερμανικά. Η δόκτωρ Αγγέλικα Ποθ Μέγκελε Διευθύντρια Πολιτικής για το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών και τέλος ο κύριος Πασκάλ Γκαρέλ, ε, Γενικός Διευθυντής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Νοσοκομείων και Παροχής Υγείας. Έχει ο καθένας 5 λεπτά. Να δώσω λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Μόμπεργκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σήμερα το πρωί γιατί εκτιμούμε το ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις απόψεις μας για το ζήτημα αυτό. Οι αρχές στη Σουηδία προσπαθούν ε, μέσω των υποχρεώσεων που προβλέπει οδηγία να καλύψουν και τις δικές μας τις αρχές τις κρατικές και τις περιφοριακές. Έχουμε 27 τέτοιου τύπου δομές στην Σουηδία. Άρα η πρόταση θα έχει σοβαρές συνέπειες για μας. Προφανώς συμμεριζόμαστε το περιεχόμενο της πρότασης, δηλαδή οι κρατικές αρχές θα πρέπει να πληρώνουν τις, ε, τους λογαριασμούς τους, όπως προβλέπουν οι υποχρεώσεις τους. Απλώς εδώ υπάρχει μια σειρά από σκέψεις για το πώς θα μπορούσαμε να, δώσουμε, να βάλουμε τέρμα στις καθυστερήσει των πληρωμών και τι διορθώσει μπορούμε να κάνουμε. Λόγω χάρη θα μπορούσε να υπάρξει προθεσμία των 30 ημερών που να είναι υποχρεωτική. Όμως αυτό που θα ήθελα να κάνω με τη σημερινή μου παρέμβαση είναι να επικεντρωθώ στις προτάσεις που έχουμε μπροστά μας, εφόσον μιλάμε για το 5% μεταξύ άλλων για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Αυτό εμπίπτει στο άρθρο 5 και υπάρχουν δύο διαφορετικών ειδών κυρώσεις που θα επιβληθούν στις κρατικές αρχές όπως οι πληρωμές με τόκο Και το άρθρο 4 που προβλέπει ότι οι κρατικές αρχές πρέπει να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους. Πρέπει λοιπόν <clears throat> να τεθούν εδώ κάποια όρια, κάποιες κόκκινες γραμμές μας απασχολούν οι δυσκολίες που προκύπτουν και διάφορα, τα διάφορα εμπόδια. Η πρόταση μπορεί να γίνει αντιπαραγωγική γιατί στόχος είναι απλώ οι κρατικέ αρχές εγκαίρω να πληρώνουν, να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους, βάσει των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Είναι ένας στόχος αξιοέπαινο και απόλυτα κατανοητός όμως. Το 5% εφόσον ισχύει από την πρώτη μόλις πληρωμή, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το πρόβλημα ίσως να διωγγωθεί. Διότι οι κρατικέ αρχέ. μπορεί να δυσκολευτούν να καταβάλουν τις πληρωμές τους σε 10 ή σε 100 ημέρες. Δεν νομίζω ότι αυτό το μέρος της πρότασης έχει μελετηθεί επαρκώς, διότι εδώ, εάν δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κάποιου μορφής κύρωση, πρέπει να δούμε το, το ποσό στην αρχική του φάση και το κατά πόσο θα μπορούσε να αυξάνεται σταδιακά. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, θα υπάρξει πρόβλημα με την υλοποίηση της πρότασης. Ο ορισμός των δημόσιων αρχών, των κρατικών αρχών, λόγου χάρη. Πώς θα συνδυαστεί με το ιδιωτικό δίκαιο, τις ανώνυμες εταιρείες. Και αυτές δεν επηρεαστούν από το άρθρο 5. και την επιβολή του ποσοστού του 5%. Κάποιες εταιρείες μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσχέρειες ως προς τις δυνατότητες ανταγωνιστικότητάς τους και ανταγωνισμού τους. Διότι πολλές φορές λειτουργούν στην ελεύθερη αγορά και στην εσωτερική αγορά σε συνδυασμό με άλλες εταιρείες. Όπως είπα ευθύ εξ αρχής, οι δημόσιες αρχές προφανώς δεν να καλύπτουν τους λογαριασμούς τους. Απλώς να τους καλύπτουν εγκαίρως. Συμμεριζόμαστε απολύτως λοιπόν την ε, φιλοσοφία που κινεί όλη αυτή την πρόταση, όμως για να ανακεφαλαιώσω πιστεύουμε ότι το 5% από την πρώτη μέρα όπου αρχίζει να τρέχει η προθεσμία δεν είναι ορθό. Δεν είναι ορθό γιατί είναι πολύ υψηλό ως ποσοστό. Μιλάμε για το 5% του ποσού του λογαριασμού από την πρώτη ημέρα, ενώ ήδη έχει καθυστερήσει η πληρωμή. Λοιπόν, πρέπει κανείς να σταθμίσει κατά πόσον το 5% θα είναι ίσως το τελικό ποσοστό στο οποίο θα φτάσει κανείς μετά από τις ε, διάφορες καθυστερήσεις, το πέρασμα των διαφόρων ημερών καθυστέρησης, θα μπορούσε εδώ να γίνει ίσως μια καλύτερη πρόταση. Καλύτερο θα ήταν, ας πούμε, να επιβάλλουμε τόκους, ε, τόκους ως κυρώσεις και ίσως διαδοχικά να αυξάναμε τους τόκους με το πέρασμα του καιρού. Αλλά θα παραμείνω σε αυτά τα σχόλια προς στιγμή. Ευχαριστώ. Mr. Κύριος Φουνστάιν. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πολύ για την πρόσκληση. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την κυρία Βάιλερ. Εγώ είμαι εσωτερικός ελεγκτής ενός Δήμου. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε μια ομάδα σε ομοσπονδιακό επίπεδο που επεξεργάζεται τις σχετικές διατάξεις, γι' αυτό και προσεκλήθηνε εδώ πέρα. Ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι στην επαρχία του Όρτενα, όπου συνορεύει άμεσα με το Στρασβούργο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν συμβαίνει το εξής. Εμείς πληρώνουμε από την στιγμή την οποία θα λάβουμε ένα ελέγξιμο τιμολόγιο. Κατά την άποψή μου λοιπόν υπάρχουν δέκα λόγοι που είναι κατά της νέας διατύπωσης αυτής της οδηγίας. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση ε, και εδώ πέρα ε, εγώ μπορώ να σας πω πως ε, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και μιλάω από την επαγγελματική μου εμπειρία στην οποία θα είχαμε καταλήξει σε ανετιολόγητες επιβολές του 5% γιατί ακριβώς πρέπει να ελέγξει ο Δήμος πριν πληρώσει οτιδήποτε. Μπορώ να σας πω επίσης περιπτώσεις οποίες μια εταιρεία παρέδωσε έναν εξοπλισμό σε τμήματα στην, ε, στον Δήμο. Ε, τελικά καταλήξαμε στα δικαστήρια και βεβαίως ο κίνδυνος θα ήταν ότι όσο εκκρεμούσε αυτή η διαδικασία θα ήταν υποχρεωμένη, να, θα ήταν υποχρεωμένη η επαρχία μας να πληρώνει. Τρίτον, και σημαντικότερον μιλάμε για χρήματα των φορολογουμένων τα οποία διαχειρίζονται οι Δήμοι, οπότε οφείλουν να κάνουν πλήρη έλεγχο πριν αποδώσουν οποιαδήποτε χρήματα Επίση δεν πρέπει να ξεχνάτε πώ μιλάμε για συμβόλαια τα οποία πηγαίνουν στην περιοχή. Στη συγκεκριμένη, να μιλήσω για τη συγκεκριμένη επαρχία του Όρτεν, 75% των δημοσίων συμβάσεων πηγαίνουν σε τοπικέ επιχειρήσει, οπότε εάν βλαφθεί τελικά ο προπολογισμό τη επαρχία θα βλαφθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και οι θέσει εργασία των τόπων μα. Επίση, το να δημιουργηθεί μία δυσπιστία θα δημιουργούσε βεβαίως και πίεση και μέσω του τύπου και δημοτικών συμβουλίων και λοιπόν αρχών οποίο βεβαίως κανείς δήμαρχος δεν θα μπορούσε να ανοιχθεί κατόπιν. Εάν δεν ε, ακολουθεί η... ο πλήρως έλεγχος δεν θα μπορέσουμε να έχουμε βεβαίως ε, ανάκτηση αχρεωστήτως ε, καταβληθέντων. Τέλος, ε, και οι ίδιες οι επιχειρήσεις ορισμένες φορές ε, φταίνε, διαπιστώνουμε πάρα πολύ συχνά στην πράξη πως δεν υποβάλλουν πλήρως τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλλουν για να πληρωθούν ή τα υποβάλλουν με μεγάλες καθερίσκα, το οποίο δημιουργεί και σε εμάς φόρτο εργασίας. Μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένο έργο κατασκευής δρόμου, όπου είχαμε αποστολή τιμολογίου 31 Δεκάτου 2006 και ξεκίνησε έφυγε αυτό το έγγραφο, μάλλον είχε συνταχθεί 31 Δεκάτου 2006, βγήκε από την εταιρεία 28 Πρώτου 2009 και πληρώθηκε εμάς 25 Τρίτου 2009. Δηλαδή εμείς εάν καθυστερούσαμε να πληρώσουμε πέρα από τις 30 ε, ημέρες θα έπρεπε να πληρώσουμε το 5% και η εταιρεία για να μας στείλει ένα τιμολόγιο έκανε δύο χρόνια. Βλέπετε λοιπόν πως και η διαχείριση των απαιτήσεων εντός των ίδιων των εταιριών ε, πάσχει ορισμένες φορές. τον, ο δημόσιος τομέας συχνά έχει και αυτός προβλήματα ρευστότητας κάτι το οποίο αποδεικνύεται εύκολα, δεν χρειάζεται να σου το πω και θα επιδεινωθούν αυτά με αυτήν την οδηγία και δέκατο και τελευταίο, αυτό το 5% θα έπρεπε να υπολογιστεί άμεσα στο κόστος, το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα είχαμε λιγότερα έργα τα οποία θα γίνονταν. Σύμφωνα λοιπόν με το γερμανικό δίκαιο, δεν θα επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες, έχουμε δοκιμασμένες ε, διαδικασίες οι οποίε είναι και υποχρεωτικές όπως σα είπα από την πλευρά του ελέγχου για να μπορέσει να εκταμείευσει ε, χρήματα το δημόσιο οπότε εγώ δεν νομίζω πως ε, θα μας οφειλήσει πάρα πολύ όπως και οπωσδήποτε αυτό το επίπεδο πρέπει να σημαίνει να υπάρξει διαφορετική μεταχείριση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι θα προκύψουν ερωτήσεις από αυτά τα οποία μας είπατε κατόπιν η κυρία Μέγκελε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια για την ε, πρόσκληση που απευθύνεται στην ε, Ένωσή μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Μπορώ να βασιστώ ευτυχώς σε αυτά τα οποία είπαν οι δύο προλαλήσαντες θα ήθελα ως εκπρόσωπος της Ένωσής μας που εκπροσωπεί 30, συνδέσμους από 37 χώρες να αναφέρω τα πολιτικά επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν από τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά δηλαδή την κρίση και την κατάσταση στις επιχειρήσεις ισχύουν βεβαίως και για τους Δήμους. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, μειώνονται οι φόροι, τα έσοδα Δηλαδή είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε και ταυτόχρονα αυξάνονται τα έξοδα όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές, οπότε βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και οι Δήμοι. Και αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες στο να βρουν και πιστώσεις. Βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση με τις ιδιωτικές ε, επιχειρήσεις. Γι' αυτό θεωρούμε και εμείς πως ε, δεν είναι σωστό ο ε, δημόσιος τομέας να τιμωρείται αυστηρότερα ε, από ότι ο ιδιωτικός. Εδώ πέρα θα θέλαμε να επικαλεστούμε την αρχή της ίσης μεταχείρισης καθώς Οπωσδήποτε οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εξαρτώνται πάρα πολύ από τα εμβάσματα των, ε, του, της κεντρικής διοίκησης και αντιμετωπίζουν και αυτή η καθυστερήση σε αυτό τον ε, τομέα. Επίσης υπάρχουν και προβλήματα πληρωμών από την ε, Ευρώπη. Πάρα πολλά κράτη-μέλη, ειδικά νέα κράτη-μέλη, εξαρτώνται πάρα πολύ από τις ε, πληρωμές του Ευρωπαϊκού Διαρθρωτικού Ταμείου, παραδείγματος χάρη, και οι ε, προθεσμίες αυτές των 30 ημερών θα έπρεπε να εφαρμοστούν είτε και στο Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο, αλλιώς θα οδηγούσαν σε μια κατάσταση αδύνατη πραγματικά για το επίπεδο της οπτικής αυτοδιοίκησης. Τώρα όσον αφορά το πακέτο αυτό της ε, ανάκαμψης ε, και το τι γίνεται σε επίπεδο Δήμου, νομίζω τα ανέφερε και ο κύριος Πφούντσταϊν το τι συμβαίνει. Μιλάμε για χρήμα του φορολογούμενου που πρέπει να ελεγχθεί πάρα πολύ προσεκτικά πριν εκταμιευθεί και υπάρχουν και πολλοί λεπτομερείς κανονισμοί που πρέπει να τηρηθούν και αυτό είναι οπωσδήποτε προς το κοινό συμφέρον, προς το συμφέρον των φορολογουμένων. Εγώ βρήκα ενδιαφέρουσα μια πτυχή που αναφέρει η κυρία Βάιλερ στο εγγραφό της και διάφοροι άλλοι προελίσσαντες. Είναι οπωσδήποτε σημαντικό πως ε, τα προτινόμενα μέτρα θα συμπληρωθούν από κάποιες ε, διατάξεις ε, και από εκπαίδευση, από ναι, ξεκαθάρισμα της όλης διαδικασίας, δηλαδή να μην έχουμε μόνο μαστίγιο, αν θέλετε, αλλά και κάποιο καρότο ειδικά έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην διαδικασία αυτή και να υποβάλουν και σωστά και έγκαιρα και γρήγορα τα... τις απαιτήσει πληρωμών. Μία άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή του εγγράφου της ε, κυρίας Βάιλερ. Μιλάτε για την αρχή εδώ πέρα του να κατονομάζονται οι οφιλέτες. Σημαντικό είναι νομίζω να τονίσουμε πως ε, και οι δήμοι στην περίπτωσή μας αλλά και οι επιχειρήσεις έχουν ένα συμφέρον για έναν, ε, προς ένα εξορθολογισμό του συστήματος και να έχουν και μια καλή επιχειρηματική σχέση. Κανέναν δεν συμφέρει αυτή η κατάσταση. Γιατί αυτό έχει βεβαίως και αρνητικό αντίκτυπο και στον Δήμο, εάν θεωρείται κακοπληρωτής. Τώρα σύντομα για το 5% για το ποσό αυτό που αναφέρατε, το ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του 5% ε, συνολικά, να ισχύσει δηλαδή αδιακρίτως. Θα πρέπει λίγο να το δείτε έτσι με κάποια περισσότερη φαντασία, ειδικά γιατί το 5% αν ισχύσει ανεξαρτήτως ε, του συνολικού ποσού, δεν το βρίσκουμε πάρα πολύ σωστό. Θα θέλαμε ε, να το δείτε έτσι λίγο με περισσότερη φαντασία το τι δηλαδή θα έπρεπε να γίνει και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Τώρα συγκεκριμένα για, τα, για τις 30 ημέρες μόνο για τον δημόσιο τομέα και αυτό δεν το βρίσκουμε σωστό. Ε, ενδιαφέρον ε, ήταν αυτό το οποίο ακούστηκε, δηλαδή 60 ημέρες για όλους, ιδιώτες και δημόσιο. Νομίζω αυτό ήταν κάτι που θα έπρεπε να το σκεφτείτε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος ο κύριος Γκάρελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Βάιλερ η οποία μας εκάλεσε. Ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό για ε, τον κλάδο των ε, ε, ξενοδοχείων. Ε, εκπροσωπούν το 9% του τζίρου του πλούτου στην ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι σημαντικό. Και άρα είναι σημαντικό να ακουστεί η φωνή μας. Η, η, ο φορέας μας ε, εκπροσωπούνται εδώ και οι υπηρεσίες υγείας, νοσοκομεία κλπ. 32 φορείς από 27 χώρες και αναχώρα. Επομένως, εκπροσωπούμε ε, ιδρύματα, ε, κερδοσκοπικά ή όχι. Πολλές φορές εκτός από νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες υγείας. Κάποιες τώρα διευκρινήσεις όσον αφορά τα νοσοκομεία. Έχουμε κάποια κρατικά νοσοκομεία ε, και όλα και λιγότερα νοσοκομεία είναι κρατικά, οπότε και εμπλέκονται όλο ένα και λιγότερες ε, κρατικές αρχές. Πολλές φορές πάντως είναι δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πάντως, το πιο σημαντικό είναι να εξετάσουμε από πού προέρχονται οι πόροι. Κατά πόσον είναι επομένως δημόσιοι οι πόροι που χρησιμοποιούνται. Πολλές φορές επομένως υπάρχει ένα φαινόμενο σώρευσης και πολλές φορές οι χρηματοδότες είναι το κράτος, τοπικές αρχές ή φορείς της κοινωνικής πρόνοιας. Και έχουμε πολλές φορές πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα όπως αναφέρθηκε σήμερα σε κάποιες χώρες ή άλλες. Δεν υπάρχουν προβλήματα καθυστέρησης πληρωμών στον κλάδο μας. Επομένω δεν θα πρέπει να υποτιμάτε το πρόβλημα κυρίως όσον αφορά τις ΜΜΕ. Έχουμε δεδομένη αυτή την έκθεση που ανέθεσε η Επιτροπή. Ιταλία, Τσεχία, Πορτογαλία και Μάλτα είναι ακραίες περιπτώσεις. Όμως είναι απογοητευτική ανάλυση διότι πολλά από αυτά που ελέγχθησαν ήταν επιφανειακά. Πολλέ φορέ έχουμε πάνω από δεκαετία καθυστέρησης ε, και ήταν, η, η ανάλυση αυτή βασίστηκε στο ίντερνετ, σε άρθρα εφημερίδων και δεν αναφέρεται καθόλου τις τόσε χώρε που έχουν λύσει το πρόβλημα. Δεν είμαι βέβαιος πάντω ότι εμεί, το δικό μα κλάδο, έχουμε καλέ επιδόσεις. Και δεν ξέρω καν αν η λύση προτείνεται αρκεί για τι τέσσερι προαναφερθήσει χώρε. Ομόφωνα θεωρούμε ότι υπάρχει δυσαναλογία σε κάποια σημεία στην πρόταση τη επιτροπή. Αυτό το 5% πρώτα-πρώτα. Δεν έχει ακόμα λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα. Δεν θα λυθεί με το 5%. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το 5% έρχεται να προσθεθεί στο νόμιμο επιτόκιο. Για μας επομένως αυτό είναι δυσανάλογο. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο θεωρούμε ότι εδώ γίνεται δυσμενής διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είπαμε ότι πολλές φορές είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Και εδώ ανακύπτει το πρόβλημα και για αυτό το 5%. Γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν φτιάξει ανταγωνισμό μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού κλάδου. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αδικίες βάρος ενός των δύο ανταγωνιστών. Επίσης θεωρούμε ότι αυτό το 1% σχετικά αφορά τις ε, μεγάλες ε, συμβάσεις και αυτό είναι δυσανάλογο. Άρα, θεωρούμε ότι αυτό το 5% θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί το 1% με κάποιο σταθερό συντελεστή όπως γίνεται και για τις μικρότερες συμβάσεις. Εν κατακλείδη, έχουμε μια μελέτη του MIT, πολύ πρόσφατη, μόλις τώρα βγήκε. Εκεί υπάρχουν εύστοχες λύσεις για να λυθούν τα προβλήματα και για ε, τις χώρες που βρίσκονται σε ακραία κατάσταση και για τις άλλες. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε εμείς, λέει ο κύριος Χάρμπορ. Τι να σας πω, ο κύριος Μπασάνη μας είπε κάποια στοιχεία την Ιταλία που ενώ μας είναι το 2009, εμένα μου φάνηκαν ότι είναι μια δεκαετία μπαγιάτικα. Τέλος πάντων. Για να δούμε τώρα ποιοι έχουν ζητήσει το λόγο. Για να μιλήσουν και οι βουλευτές. Η κυρία Βάλια πρώτα από τα φίλη να απαντήσει κάποιες ε, ερωτήσεις. Κατόπιν έχουμε Γκέμπχαρτ, Σβάρμπερ και Ριζόρντι. Διόν, που είναι ο σκιοδησηγητής που και αυτός πρέπει να λάβει το λόγο. Κατόπιν έχουμε Άριας, Μάντερς και άλλους. Α, και, ο κύριος Κρότσμαν έχει ζητήσει το λόγο. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουν οι το λόγο. Ποιος άλλος είναι? Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να λάβετε το λόγο. Να είσαστε όμως σύντομοι γιατί θέλουμε και η Επιτροπή να λάβει το λόγο. Κυρία Βάιλερ, παρακαλούμε να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Και κατόπιν κυρία Μπιέγκχαρτ. Να πω κάποια πράγματα για τα μαστίγια και τα καρότα που ακούστηκαν. Επειδή ετέθη το ζήτημα να ξεκαθαρίσω κάτι, είναι σημαντικό για όλους μας και για εσάς που είστε οι ειδικοί, ε, αυτή η οδηγία θα ισχύσει και για την Κομισιόν. Γιατί είχαμε ε, φοβηθεί όταν διαπιστώσαμε ότι δεν ίσχυε στο παρελθόν για την Κομισιόν. Στο μέλλον θα ισχύσει πάντως. Ευχαριστώ. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί γνωρίζουμε και το τι σημαίνουν οι καθυστερήσεις ε, όταν καθυστερεί η Κομισιόν να πληρώσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Λοιπόν τώρα, επειδή πιέζει ο χρόνος, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Μπάτερς και στον κύριο Φουντστάιν. Άκουσα πάρα πολλά πράγματα για την αρχή αυτή της ελευθερίας συμβάσεων γιατί ισχύει αυτή για τις επιχειρήσεις αλλά όχι για τον δημόσιο τομέα ή για τις δημόσιες προμήθειες. γιατί δεν θα πρέπει να ισχύει για τον δημόσιο τομέα, γιατί αυτή η άνηση μεταχείριση. Δεύτερον, κύριε Μπάτερς, μας είπατε πως ε, είναι μη αναλογικό το να πούμε ότι είναι 5% κατά αποκοπήν. Ε, δεν μας είπατε όμως συγκεκριμένα τι εννοείτε, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και προς τον κύριο Μπορσάνη και προς την κυρία Ποτ Μέγκελε να ρωτήσω το εξής ε, όσον αφορά τον τομέα της υγείας. Μας είπε ο κύριος ε, Μπορσάνη τρομακτικά πράγματα για τον τομέα της υγείας, αλλά πολύ γενικά, χωρίς διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εδώ πέρα. Υπάρχουν διαφορές. Δεν υπάρχουν, θα θέλαμε να το μάθουμε. Και επίσης ε, πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα κράτη-μέλη όλα, όχι μόνο για την ε, Ιταλία. Υπάρχουν 27 κράτη-μέλη και όχι μόνο ένα, οπότε θα ήθελα κάποιες ε, πληροφορίες και με συγχωρείτε που είναι τόσο πολλές οι ερωτήσεις μου, είναι ακόμη περισσότερες, αλλά σταματήσω εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα στην γνωμοδότηση της ΟΕΑΠΜΕ πως η Κομισιόν αρνήθηκε να δει το ζήτημα του B2C, επιχειρήσεις προς καταναλωτές. Γιατί ε, αρνήθηκε η Κομισιόν να δώσει τέτοιες ε, πληροφορίες όταν ένας ευρωπαϊκός, μια ευρωπαϊκή οργάνωση εδώ πέρα λέει πως υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα μπορούσε να ρωτήσει η Κομισιόν ε, τους ενδιαφερομένους γιατί δεν το έκανε. Υπάρχουν και άλλε ερωτήσει προ την Επιτροπή. Θα τι ακούσουμε αργότερα. κύριο Σφάλμπ. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Βάιλερ, την εισηγήτρια για την πολύ καλή αυτή προετοιμασία της σημερινής ακρόασης πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι παρεμβάσεις. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με αυτό το οποίο τελείωσε η κυρία Γκέπχαρτ. Πιστεύω πράγματι πως το να κατανομάζουμε ε, και να ντροπιάζουμε είναι ε, λογικό, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο στην Ιταλία, δεν αφορά καθόλου μόνο την Ιταλία. Όσον αφορά δε τον τομέα της υγείας. Ξέρω πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ακριβώς κυρία Βάιλερ, που από την Ελλάδα δεν έχουν λάβει χρόνια καθόλου χρήματα. Να μην μιλήσουμε μόνο για την Ιταλία, είναι άδικο. Και θα ήθελα να πω επίσης πως το πρόβλημα αυτό το οποίο πάλι τύχθηκε σήμερα για τα πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία ακόμα εγκρεμούν τα οποία ανέφερε βεβαίως η Κομισιόν στην ε, μελέτη αντικτύπων, και είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις ε, μικρόμεσες ε, επιχειρήσεις και κατά την άποψή μου άρα νομίζω θα έπρεπε να αφορά το ζήτημα της ε, αυτονομίας του ιδιωτικού τομέα. Οπότε δεν ξέρω εάν θα έπρεπε να προβλέψουμε γενική ακυρότητα ρητρών όταν μιλάνε για προθεσμίες πέραν των 30 ημερών μετά την παράδοση του ε, προϊόντος ή υπηρεσίας. Γιατί βεβαίως όταν ε, παραδοθεί το προϊόν ή υπηρεσία ε, είναι πληρωτέο και το τίμημα. Και ε, το να υπάρχει πρόβλημα πίστοση μετά δεν έχει καμία σχέση με τον ε, επιχειρηματία. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω συγκεκριμένα εδώ πέρα την άποψη του κ. Χέντριξ. Τώρα για τον κύριο Μπορζάνη μπορεί να μα ε, διευκρινίσει γιατί θεωρεί πω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει πρέπει να έχουν διαφορετική μεταχείριση από τη βιομηχανία. Και προ τον κύριο Πφούντστάιν το εξή ερώτημα. Ποιο θεωρεί πω θα πρέπει να είναι ο προπολογισμό των έργων και των δημοσίων συμβάσεων στο μέλλον, ε, εάν είναι να συνυπολογίσουμε αυτό το 5% την ρήτρα αυτή, ε, εάν δηλαδή γίνει πραγματικότητα αυτή η πρόταση, πώς θα κινηθείτε εσείς ή θα οδηγηθούμε όντως σε αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή να μειωθεί ο όγκος των ε, έργων των, δημοσίων προμηθειών. Κύριο, κύριος Μπουζόη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πρόταση σοβαρότατη η οποία θα έχει μεγάλο αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις. Και δεν μιλώ μόνο για τις μικρομεσαίες, αλλά και για τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες προσλαμβάνουν χιλιάδες Ευρωπαίους εργαζομένους και επηρεάζουν τον προπολογισμό των κρατών μελών και τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό, την υγεία και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όσους εκπροσωπούν τις ε, δημόσιες αρχές είναι το εξής. Δεν νομίζω ότι η πρόταση αυτή θα επιβάλλει πειθαρχία στις δημόσιες αρχές. Πιστεύουν λοιπόν αυτοί οι εκπρόσωποι ότι, ότι θα αλλάξει κάτι στις καθυστερήσεις των πληρωμών και κύριε Φιονστάιν, εάν οι πολίτες πληρώνουν τους φόρους τους, εάν μάλλον δεν πληρώνουν τους φόρους τους ε, εγκαίρως, ε, τους επιβάλλονται αμέσως πρόστιμα και υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες επιπαραβάσει. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν θα υποχρεωθούν να συμμορφωθούν με αυτές τις υποχρεώσεις. Γιατί να μην υπάρχουν αναλογοί κανόνες. Τέσσερα κράτη-μέλη έχουν δυσκολίες ε, καταβολής των πληρωμών εγκαίρως. Ξέρω πολλές ε, φαρμακευτικές εταιρείες ε, στην ε, Ρουμανία που θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενες να λάβουν την πληρωμή τους 208 ημέρες μετά την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο τομέας της υγείας λοιπόν είναι πολύ ευαίσθητος. Ξέρουμε ότι στην Ευρώπη είναι πολύ ισχυρό ο κρατικός τομέας και μπορεί να πιέσει τους ιδιωτικού φορείς. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχουν εξαιρέσει. Εάν οριστούν 30 ημέρε, θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτή την προθεσμία. Ο καθένα θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τι εξαιρέσει εφόσον προβλεφθούν. Επίση, τα πρόστιμα και οι αντισταθμίσει θα πρέπει να ισχύουν αυτομάτω. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ε, αποζημίωση, αλλά αυτό δεν είναι υποχρέωση. Θα βρεθούμε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου θα ζητάτε η αποζημίωση αλλά θα τους λένε οι θα, θα απειλούνται εταιρείε ότι δεν θα ξαναλάβουν άλλη σύμβαση. Δεν μπορεί να λειτουργούν λοιπόν έτσι οι αντισταθμίσεις. Θα πρέπει να είναι αυτόματες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μεταξύ των συντονιστών τώρα. Νομίζω ότι έχω πολλούς που θέλουν να μιλήσουν, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και τους εισηγητές. Εφόσον έχουμε αυτό το υπέροχο τεχνολογικό μέσο, θα Σα βάλω και ένα χρονόμετρο για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα περβείτε τα δύο λεπτά, ώστε να έχουν άφθονο χρόνο και η Επιτροπή και οι υπόλοιποι παρεμβαίνοντε. Έχω πολλούς ομιλητές και κλείνω τον κατάλογο ομιλητών με τα ονόματα που σας ανέφερα. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και με συγχωρείτε που έχασα ένα κομμάτι, αλλά ευτυχώ έχω μιλήσει διμερό με κάποιε από αυτέ τι οργανώσει, οπότε έχω από αυτέ τι πληροφορίε. Έχω δύο-τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα έγινε μια συζήτηση για το εύρος ε, εδώ πέρα. Πράγματι είναι ουσιαστικό, εγώ συμφωνώ με το ερώτημα της κυρίας Γκέπχαρτ γιατί είναι διαφορετική η ελευθερία συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών και όταν εμπλέκεται το δημόσιο και πράγματι θα ήθελα να ακούσω και αυτό το επιχείρημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι πράγματι είναι λογικό ότι είναι τελείως διαφορετική η σχέση της ισχύω μεταξύ της μεγάλης επιχείρησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά βεβαίως το ίδιο ισχύει και για το κράτος και τους λοιπούς ε, συναλλασσόμενους. Οπότε το ερώτημά μου είναι εδώ πέρα ποιες είναι οι σοβαρές ε, συνέπειες εάν το επεκτείνουμε και στις ε, ε, συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Δεύτερον, μιλήσατε για τις τοπικές αρχές. Μπορώ να σας πω πως στην Ολλανδία έχουμε νομοθεσία 30 ημερών, λειτουργεί, δεν έχει ξεσπάσει καμία επανάσταση, καμία εξέγερση. Εξακολουθούν να εκπληρώνονται οι λειτουργίες των τοπικών αρχών δεν ξέρω αν έχετε επαφές με συναδέλφους ε, σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω γιατί σε ορισμένες χώρες γίνεται και σε άλλες όχι. Δεν είμαι πολύ πεπισμένος για αυτό το επιχείρημα του ότι θα παραλύσουν τα πάντα με τις 30 ε, ημέρες. Μιλάμε για 30 ημέρες από την παράδοση του παραδοτέου προϊόντος ή υπηρεσίας. Τέλος, ε, είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση το ότι λέμε ε, είτε 90 ημέρες είτε ένα χρόνο μετά εγώ πρέπει να πληρώσω 5% κατά αποκοπή. Αυτό μου φαίνεται κάπως ε, αυθαίρετε. Θα ήταν καλύτερο να πούμε πως θα έχουμε συγκεκριμένη προσάυξηση ε, επί του τόκου αντί για το συγκεκριμένο 5% και όσο βεβαίω παρατείνεται η καθυστέρηση να ανεβαίνει αυτό το ποστό. Σας φαίνεται καλύτερο αυτό το σενάριο. και θα το λέω Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις ε, προς τον κύριο Πφούντσταϊν. Είπατε ως δήλωση πως πάντα στην ώρα τους πληρώνει το, πληρώνει το δημόσιο και μετά λέτε πως πρέπει να συνυπολογίσουμε και το 5%. Ε, εδώ πέρα μου φαίνεται πως ε, υπάρχει κάποια αντίφαση. Αν πληρώνετε πάντα στην ώρα σας δεν έχετε να, φοβάτε, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Κατόπιν. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την οδηγία. Μιλάμε για 30 ημέρες μετά την λήψη τιμολογίου ή απέτηση πληρωμής. Δεν μιλάμε για 30 ημέρες μετά την παράδοση του έργου. Εάν σας στείλουν το τιμολόγιο τρία χρόνια μετά, από εκείνη τη στιγμή μιλάμε 30 ημέρες. Είναι σημαντικό αυτό νομίζω. Και βεβαίως ε, είναι γνωστό, ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, γνωρίζουν πάντα τι γίνεται, έχουν θέμα με την ρευστότητα, οπότε σας παρακαλώ διαβάστε τι γράφει εδώ πέρα. Είναι 30 ημέρες μετά τη λήψη του τιμολογίου ή την απέτηση πληρωμής. Κύριε Ρούλερ, ε, και εγώ στο ίδιο σημείο φοβάμαι πως αυτή η οδηγία δεν θα έχει το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους σκιώδεις και τους συντονιστές να έχουμε αρκετό χρόνο για να την ανασυντάξουμε, να την ξαναγράψουμε. Δεν νομίζω πως έκανε καλή δουλειά εδώ πέρα η Κομισιόν, μιλάμε για τις 30 ημέρες, αλλά εάν δούμε ακριβώς 30 ημέρες. Υπάρχουν πάρα πολλές εξαιρέσει που θα οδηγήσουν ακριβώς στο ότι χώρε όπως η Ελλάδα και η Ιταλία πάλι θα καταφέρουν να βρουν ε, κάποιον τρόπο να το παρακάψουν και οι υπόλοιποι απλά θα είναι πιο ε, θα στριμωχτούν ακόμη περισσότερο. Οπότε, 60 ημέρες για όλους, αντί να βρούμε όλες αυτές τις εξαιρέσεις. Και πρέπει να σκεφτούμε τι προσφέρουν οι εξαιρέσεις. Τι μας προσφέρει αυτή η μη καθαρή κατάσταση και θα οδηγήσει στις χώρες στις οποίες ούτως ή άλλως δεν ήταν πολύ ικανοποιητικά τα πράγματα ε, στο να χειροτερέψει ακόμα η κατάσταση και να έχουμε εδώ πέρα έναν τίγρη χωρίς Το ίδιο και για το 5% ακούγεται πολύ αυστηρό, ακούγεται πολύ σκληρό, αλλά στην πραγματικότητα έχει δίκιο ο κύριος Πφούντσταϊν. Αν σκεφτούμε π.χ. πάλι την Ελλάδα και τα γνωστά προβλήματα, Τίποτα. Θα, θα συνυπολογιστεί. Δεν, ε, ε, δεν, δεν θα έχει κανένα όφελος. Γι' αυτό σωστό ήταν αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος νομίζω. Πρέπει να πάμε προ αυτή την ε, κατεύθυνση που είπε ο κύριο Γιόγκ. Και τέλος ένα ερώτημα προς την ε, Κομισιόν. Γιατί δεν είχε όλες τις οδηγίες που είχαν συμπεριληφθεί αρχικά, η 2004-17. Γιατί περιορίσατε εδώ πέρα το πεδίο εφαρμογής. Ευχαριστώ για τα πολύ σαφή αυτά σημεία. Οπωσδήποτε κανείς εδώ πέρα δεν θέλει ε, ένα τίγρη χωρίς δόντια, όπως είπατε. Λοιπόν, κύριος Κοσνέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάτι θα πρέπει να γίνει ούτως ώστε να μπορέσουμε να εμπλέξουμε δήμους και κοινότητες. Θα πρέπει να απευθυνθούμε και σε αυτούς και να ακούγεται μεταφράζονται αυτό που λέω ναι, ναι. Επομένως θα πρέπει να απευθυνθούμε στους φορείς το, της ε, αυτοδιοίκησης και να επικοινωνήσουμε, να διαβουλευτούμε με αυτούς τους φορείς, διότι κατά τη γνώμη μου παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτούς, αυτούς που έχουν τα δικά τους προβλήματα και συνάπτουν και συμβάσεις μεταξύ τους. Επομένως, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό το 5% αντί να λύσει το πρόβλημα, το δημιουργεί ε, όσον αφορά μια κύρωση σε περίπτωση υπερημερίας. Προσοχή, μήπως το δημιουργήσουμε προβλήματα όπως διαφθορά κλπ. Συνήθω, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει πρόβλημα αυτές τις 30 μέρες. Δυστυχώς το πρόβλημα ανακύπτει όταν έχουμε συγχρηματοδότηση με την ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση οι καθυστερήσει είναι πολύ μεγαλύτερε από 30 μέρες. Uh, thank you very much for your practical researches, which I think is very impressive. Πάρα πολύ ε, ουσιαστικά και που μας είπατε επόμενο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο Πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι το πρόβλημα 30, 60, 90 μέρες. Το πρόβλημα είναι κάποια χρόνια καθυστερήσεων. Άρα κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Επίσης συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Είναι κάπως απονευρωμένη αυτή η οδηγία, γιατί για να δούμε όσον αφορά τις κρατικές αρχές. Εάν θέλουμε να πούμε για κάτι το οποίο έχει συγκεκριμένα συμφωνηθεί μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη, τότε τι γίνεται όσον αφορά τις κρατικές αρχές σε περίπτωση που κάνουν κάποιο διαγωνισμό και δεν είναι θέμα πια ε, διμερούς σύμβασης. Να μας πει η Κομισιόν πώς αυτό θα το ε, θα το νομοθετήσουμε, τη σχέση δηλαδή οφειλέτη και Πιστοτή Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε για το κράτος. Εννοούμε νομικά πρόσωπα, εννοούμε μόνο το, το κράτος, τι. Τώρα όσον αφορά αυτά τα, τις δαπάνες ανέκτησης πάσα δαπάνη θα πρέπει να καλύπτεται. Ό,τι δεν καλύπτει το νομικό πρόσωπο. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στις ΜΜΕ. Άρα ο ορισμός αυτός θα πρέπει να διευκρινιστεί. Επίσης, για την ελαχίστη αποζημίωση, να δούμε τι γίνεται με αυτό τα 40 ευρώ. Σε πολλές χώρες νομίζω ότι αυτό το ποσό δεν, δεν, δεν έχει νόημα. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρος. Άριας. Μπαρνιέ, Μάντερς Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θα διαφωνήσω κατά κάποιο τρόπο με όλα όσα ακούσαμε. Να σας πω τις σκέψεις μου όσον αφορά αυτό το τρίακονταήμερο και όσον αφορά την αποζημίωση του 5%. Αυτή η προθεσμία είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο καλώς έχει, αλλά όσον αφορά αυτή την αποζημίωση για κάποια μήμη δεν αποτελεί λύση. Γιατί η ΜΜΕ θέλει χρήματα, πρέπει να, να πάρει κάποια λεφτά. Επομένως, όσον αφορά τη σύμβαση με το κράτος, μάλλον κάποια ταμιακή διευκόλυνση, κάποιο χρηματοδοτικό μέσο από πλευρά του κράτου θα βοηθούσε περισσότερο τη ΜΜΕ. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο και πολύ πιο απλό αυτό. Και βέβαια πολύ λιγότερο γραφειοκρατικό. Γιατί πάντοτε ζημιωμένε βγαίνουν οι ΜΜΕ από τέτοιε συμβάσει. Για τον τη κοφίντου, βεβαίω θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ μικρών και μεγάλων ε, επιχειρήσεων. Ε, γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο και όταν έχουμε μια, μια μεγάλη μια μικρή επιχείρηση, ε, πιο μικρή είναι αυτή η οποία βγαίνει ζημιωμένη. Μιλούμε τώρα για ιδιωτική σύμβαση. Άρα είμαι υπέρ της ελευθερίας των συμβάσεων. Όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη για την ομοθεσία μας ότι δεν είναι σε θέση ισχύω. Είναι η πλευρά η ΜΜΕ σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άριας. Λέει ο πρόεδρος. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εδώ τον κύριο Μπαρνία. Και επίσης συγχαρητήρια όσον αφορά την υποψηφιότητα για τη θέση του Επιτρόπου για τη Γαλλία. Μαλά με μεγάλη μας χαρά. Σας έχουμε εδώ να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ για καλά σας λόγια, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι, βέβαια και για μένα είναι πάρα πολύ ευχαριστώ να βρίσκομαι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να γίνει, εδώ γείτονε θα είμαστε. Θα συνεργαζόμαστε όπως κάναμε πάντα. Πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Μπράβο που την οργανώσατε αυτή η πρακτική είναι πάρα πολύ επιζήμια. Κάνει ε, πάρα πολύ κακό στις ε, μικρές επιχειρήσεις και σε ε, συγκυρία τέτοια κρίση είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα επομένως. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια οδηγία, ένα σχέδιο οδηγίας. Και πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία ακούστηκαν εδώ Ιδίως να ευχαριστήσουμε τους ε, εμπειρογνώμονές μας για τη συμβολή τους. Να σας πω ποια σημεία θεωρώ πιο σημαντικά στο κείμενο. Το πεδίο εφαρμογή πρώτα απ' όλα. Η διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παραγωγές επιχειρήσεις έχουν τρόπο να ασκήσουν πίεση. όπως και δημοσιοφορεί, τόσο ώστε να μπορέσουν να επιβάλλουν κάποιο είδου ε, προθεσμίε από τις Όπως είπε και ο συνάδελφος ε, ε, από τη Γαλλία, θα πρέπει από το πιθανομίες να γίνουν κάποιες εξαιρέσει, κάποιες παρεκκλήσει. Για τις ε, τώρα, κύριε Βάιλερ όσον αφορά αυτή την αποζημίωση, αυτό το κόστος ανάκτησης. Θα πρέπει να έχουμε ενιαία κριτήρια ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης, δεν είμαι ο μόνος που διαφωνώ το 5% και εγώ θεωρώ ότι είναι δυσανάλογα μεγάλο αυτό το ποσό, αυτό το ποσοστό. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε ένα άλλο σύστημα. Προοδευτικό, αναλογικό, όπως θέλετε πέστε το. Ευχαριστώ. And thank you very much for respecting your speaking time. Σας ευχαριστούμε που παραμείνατε στα όρια του χρόνου ομιλίας σας. Την επόμενη φορά θα έχετε περισσότερη ελαστικότητα από πλευράς μου. Κύριε Μάντελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και εμπειρογνώμονες, διότι είναι πολύ σοβαρή αυτή η έκθεση. Εδώ ομιλούμε για, για ένα κρυφό οικονομικό σύστημα ουσιαστικά. Ένα υπόγειο σύστημα παραοικονομίας. Δεν θέλω να πω στις λεπτομέρειες, αλλά έχω δύο ερωτήσεις προς τους ειδικού. Η πρώτη είναι, Πιστεύετε ότι είναι επιθυμητό να έχετε απευθείας ένα τίτλο ώστε να μην χρειάζεται να πάτε στο δικαστήριο πριν να σας πληρώσουν τα επιπλέον 40 ευρώ ή εφόσον είναι περισσότερα περισσότερα. Και το άλλο είναι ότι όλοι οι ειδικοί και συνάδελφοί μίλησαν για την ειδική μεταχείριση και τον ιδιωτικό δημόσιο τομέα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες. Ξέρουμε ότι τα σούπερ μάρκετ πληρών, πολλούν ήδη πολύ πάνω τη τιμή του κόστου ε, προϊόντα πριν καν αρχίσει η πληρωμή του. Λοιπόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οδηγία αυτή μήπω πρέπει να γίνει κανονισμό ώστε να έχουμε ίση μεταχείριση σε όλη την Ευρώπη, διότι αν η οδηγία παραμείνει τέτοια, εφόσον μεταφερθεί στην ε, εθνική νομοθεσία θα καταλήξουμε σε 27 διαφορετικέ προσεγγίσεις. Καλό είναι να έχουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση. Θα ήθελα να ακούσω πραγματικά τι απόψει των ειδικών επ' αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η παρατήρησή σου για την συμμετοχή των τραπεζών εδώ. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον η Επιτροπή Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων θα έπρεπε ίσω να συμμετέχουν περισσότερο στη συζήτησή μα για τι διευκολύνσει που θα παρέχουν οι τράπεζε ε, ω προ το ρευστό στι δημόσιε αρχέ για την καταβολή των πληρωμών του. Ο κύριο Σάιμον, τελευταίο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα σουν σερβάντα, λέμε. Είναι αυτό βασική αρχή του δικαίου και είναι κάτι που ισχύει και για τι 27 χώρε μέλη. Γι' αυτό και για μένα δεν είναι τόσο σαφέ το γιατί θα πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αν έχουν μια παρόμοια συμπεριφορά όσον αφορά τις ε, πληρωμές τους. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα το αυτό λέει και η Κομισιόν, το ίδιο και οι υπόλοιποι. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση όταν σε μια αγορά δρά και το δημόσιο και, το, και ο ιδιωτικός ε, τομέας γιατί το πρόβλημα είναι ο ιδιωτικός. Εδώ, ε, ή ο δημόσιος μόνο. Αυτή την αιτιολόγηση θέλουμε εδώ πέρα για να μπορούμε να δούμε αν πράγματι χρειάζεται διαφορετική μεταχείριση του δημόσιου τομέα. Γιατί λοιπόν αναρωτιέμαι εγώ εδώ πέρα είναι τέτοια η αντιμετώπιση της Κομισιόν και λέει μόνο ο δημόσιος ε, τομέας όταν ξέρουμε πως υπάρχει και ανάλογη σχέση μεταξύ των μεγάλων και των μικρών εταιριών όταν είναι οι μεν ε, προμηθευτές των δε. Εάν ο στόχος μας είναι να παρεμβούμε εκεί πέρα όπου υπάρχει ανταγωνισμός δίκαιος και ελεύθερος μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα οδηγηθούμε σε μια απαράδεκτη στρέβλωση. Πρέπει να δούμε ποια είναι η βάση. Ε, γιατί προτείνει η Κομισιόν εδώ πέρα στρέβλωση της αγοράς. Νομίζω η κυρία Ρούλε εδώ πέρα με την πρόταση μιας ε, επαναδιατύπωσης της ε, οδηγίας ε, πραγματικά θα βρει πολλούς ε, να συμφωνήσουν μαζί της, μεταξύ των οποίων και εγώ. Και νομίζω, νομίζω πως κάτι τέτοιο είπε και ο κύριος Φούντσταϊν, το οποίο παρεξηγήθηκε ή δεν ακούστηκε. Δεν μιλάμε απλά για τιμολόγια. Μιλάμε για τιμολόγια τα οποία είναι ελέγξιμα και ακριβώς εδώ είναι το θέμα της ε, πληρωμής του δημοσίου. Και κάτι άλλο τεχνικό, ο διαχωρισμός μεταξύ ε, προσαυξήσεων και τόκων, γιατί βεβαίως οι προσαυξήσεις εδώ πέρα που έχουμε είναι και αυτές κατά βάση ένα είδος ε, τόκου ο οποίος έχει γίνει μια καταποκοπή πληρωμή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τη δεύτερη ομάδα υπηρεγνωμών να απαντήσει. Για να τους βοηθήσω θα τους δώσω δύο λεπτά ενδεικτικά στον καθένα για να υπάρχει χρόνος και για την Κομισιόν. Ο κύριος Μόμπερκ. Eh, ευχαριστώ το ζήτημα νομίζω ότι εξετάστη εντελεχώς. Εγώ στάθηκα στο ποσοστό του 5%. Και εγώ το ανέφερα στην εισαγωγή μου. Πολλοί μίλησαν για το ποσό αυτό. Και α, ε, υπήρξαν πολλοί που είπαν ότι το ποσοστό στην αρχή θα έπρεπε να είναι χαμηλότερο και να αυξάνεται σταδιακά. Εδώ Μιλήσαμε για τις αιτιολογήσει των πληρωμών. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και νομικά μέτρα τα οποία διησχύουν, διότι μια πληρωμή όταν δεν καταλαβ... καταβάλλεται θα πρέπει να μπορεί κανεί να καταφύγει και σε νομικά μέτρα, να μπορεί να προσφύγει σε ένα δικαστήριο. Να πάρει μια εντολή επιβολής ε, των μέτρων από το δικαστήριο. Υπάρχουν λοιπόν ένδικα μέσα για να λάβει κανείς την πληρωμή του. Τώρα όταν μιλάμε για τον ε, τομέα της, ε, τον υγειονομικό και στη Σουηδία υπάρχουν ε, πολλοί φορείς και ιδιωτικοί μεταξύ άλλων και φαίνεται η πρόταση να μην καταστά τα πράγματα πιο σαφή. Ιδίως ως προς τους δημόσιους φορείς εδώ. Διότι πηγαίνουμε πάλι στο ποσοστό αυτό του 5% το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στους ε, ε, ε, αρμόδιους να πληρώσουν μεν εγκαίρως, αλλά εάν δει κανεί ότι τα ασφάλματα είναι ανθρώπινα, θα πρέπει να ξέρουμε από πού ακριβώ θα αρχίσουμε. Κύριε Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ίσως θα έπρεπε να ξεκαθαρίσω λίγο καλύτερα. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε δύο λεπτά. Τώρα για το τι ισχύει. Ε, κοιτάξτε, για προϊόντα και υπηρεσίες έχουμε προθεσμία 30 ημερών από όταν θα έρθει σε εμάς, όπως σας είπα, ελέγξιμο τιμολόγιο και αυτή είναι η σημαντική λέξη. Δεν είναι αυτό όμως το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ συχνά στα οικοδομικά έργα. Εκεί πέρα δεν τηρείται η προθεσμία των 30 ημερών γιατί θα πρέπει εντός 18 ημερών να γίνουν οι πλήρωμες σε δόσεις και μετά να πληρωθεί το τυχόν υπόλοιπο αλλά όπως σας είπα εδώ πέρα είναι σημαντικό, όπως είπα πάλι αυτή η λέξη των ελέγξιμων ε, τέτοιων, ε, των ελέγξιμων ε, τιμολογίων, αλλά όπως σας είπα χρειάζεται και νομίζω εδώ πέρα πρέπει να μείνουμε συμβασμό των 60 ημερών, γιατί χρειάζεται ένας χρόνος και η κάθε δημόσια αργή να ελέγξει αυτά τα οποία αποστέλλονται. Κοιτάξτε τώρα, κάτι άλλο. Όταν κάνετε δημοσκοπήσεις και λένε οι επιχειρήσεις πως δεν μας πληρώνει εγκαίρως ο δημόσιος τομέας μπορεί να ήταν να απάντησε σε αυτό και η επιχείρηση η οποία σας είπα έκανε δύο χρόνια να μας στείλει το τιμολόγιο και εμείς μας το έστειλε τέλος Ιανουαρίου και πληρώσαμε Μάρτιο. Οπότε μέσα στις 60 ημέρες ήμασταν, αλλά εάν γίνει 30 ημέρες θα είχαμε και με αυτή την περίπτωση πρόβλημα για να επανέλθω σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά λοιπόν τώρα τον υπολογισμό του κόστους και το 5% εγώ θεωρώ πως θα ίσως προϋπολογίζονταν, αλλά εδώ πέρα χρησιμοποιώ υποθετική φωνή στον προϋπολογισμό, εάν τεθεί ενισχύ μια τέτοια ε, διάταξη, αλλά υποθέτω, ελπίζω πως ε, θα οδηγηθούμε σε 60 ημέρες και νομίζω πως δεν θα έχουμε προβλήματα όταν μιλάμε πάντα για ε, απαιτήσει οι οποίες μετά δεν υπόκεινται σε καμία αμφισβήτηση. Ποτ Ναι, ε, από την ε, ποιότητα των ερωτήσεων διαπιστώνω πως οι κυρίες και κύριοι εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ε, ενημερωμένες και ενημερωμένοι για τα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα εγώ να αναφερθώ σε μία συγκεκριμένη πτυχή. Βεβαίως είναι διαφορετική η κατάσταση στο κάθε mm-hmm. κράτος μέλος. Και αυτό βεβαίω οφείλεται και στο πώ εφαρμόζεται η κάθε οδηγία στο κάθε κράτο μέλο. Γνωρίζετε πω υπάρχει και η γνωστή βαθμολογία τη Κομισιόν, γιατί βεβαίω υπάρχει και η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, αλλά και η ουσιαστική εφαρμογή που είναι κάτι διαφορετικό. Και εκεί πέρα θα έπρεπε να δώσουμε βάρο στην ε, πραγματική εφαρμογή. Και βεβαίω υπάρχουν και τα καλά παραδείγματα. Όπως ξέρετε η Ολλανδία, το γνωρίζουμε και από τις ε, συναδέλφους μας, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να λειτουργήσουμε τις 30 μέρες. Σε κάποιες άλλες χώρες είναι αλλιώς η κατάσταση. Νομίζω μπορούμε να διδαχτούμε από τις βέλτιστες πρακτικές να υπάρξει μια ανταλλαγή εμπειρίας ε, δηλαδή με, τις, ε, με τους ΟΤΑ εκεί πέρα να δούμε το τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να σκεφτείτε και να σκεφτούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το τι μπορεί να ρυθμιστεί και το τι μπορεί να παραμείνει στην επικουρικότητα, ειδικά στα κράτη εκείνα μέλη στα οποία υπάρχει στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο ήδη ε, κάποιος κανόνας και υπάρχει μια καλή και δοκιμασμένη πρακτική η οποία θα έπρεπε ίσως να διατηρηθεί. Ευχαριστώ. Euh, για τον υγειονομικό τομέα, για άλλη μια φορά, πρέπει να ξεκινήσουμε από το τι μπορούμε να μάθουμε από αυτού έλυσαν το ζήτημα. Ανέφερε ο κ. Γιόγκ το παράδειγμα των κατοχωρών. Πώ τα κατάφεραν, αυτό είναι το ερώτημα. Και άλλε χώρε τα έχουν καταφέρει. Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία δηλαδή. Οι σκανδιναβικέ χώρε δεν έχουν αυτό το πρόβλημα στο υγειονομικό τομέα. Σημαντικό λοιπόν το στοιχείο. Πώ τα κατάφεραν, πώ τα κατάφεραν. Και μια σωστή παρατήρηση για την ανάλυση του τομέα τη υγεία αριθμού και αν είναι παλιό ή όχι. Ε, δεν είναι ακριβώς το 2009. Θα σας ε, παραπέμψω στην αναθεώρηση, την έκθεση αναθεώρησης για την νομοθεσία στον υγειονομικό τομέα, ε, ένα έγγραφο δεκαετίας. Και επίσης προσοχή στην, σε επιπτώσει που μπορεί να έχει το ποσοστό του 5% στις υγειονομικές μέρημνες. Δηλαδή, η προθεσμία των πληρωμών και οι εξαιρέσει μπορεί να επηρεάσουν γιατί πολλές φορές και αυτοί που δεν πληρώνουν στον υγειονομικό τομέα είναι θύματα των χρηματοδοτών, των τους. Οπότε οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη και αυτό το στοιχείο. Uh, Κοιτάζω τώρα το ρολόι μου. Και ξέρω ότι και οι πρώτοι μας εμπειρογνώμονες θα ήθελαν να είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν ξανά. Να σας δώσω από ένα λεπτό να απαντήσετε και εσείς σε μερικές από τις παρατηρήσεις που ακούσατε στο δεύτερο γύρο. Ιδίω όσα ακούσατε για τις δημόσιες αρχές. Κύριε Μπάτερς, για ένα λεπτό. Μία μόνο ερώτηση αφορούσε εμένα. Προέρχεται από την κυρία Γκέμπχαρτ και αφορά αυτό το 5%. Είπαμε για δυσαναλογία. Ίσως πιο σωστό είναι να το χαρακτηρίσουμε αυθαίρετο, όχι δυσαναλόγο. Άρα επομένως θα πρέπει να γίνει κάπως πιο δόκιμη προσαρμογή σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το ποσό. Γι' αυτό σας λέω, είναι αυθαίρετο. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τόσο μας είπαν οι εκπρόσωποι των κρατικών φορέων, ότι δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα θα παραξενθεί και όχι θα λυθεί. Άρα θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά. Βεβαίω και δεν συμφωνώ με τα επιχειρήματα των κράτηστων, θα πρέπει όντω να μην συνάπτουν συμβάσει οι κρατικοί φορεί αν νομίζουν ότι δεν μπορούν να, να, να τηρήσουν τα, τα, τα υπεσχημένα. Αυτό το οποίο ισχύει άλλωστε για τι επιχειρήσει. Πάντω να είμαστε ρεαλιστέ και να σκεφτούμε ποιε θα είναι οι συνέπειε ενό τέτοιου 5%. Κυρία Χέρινγκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι το σχολείο της κυρίας Γκέπχαρτ απευθυνόταν στην Επιτροπή, έτσι. Ωραία. Θα τονίσω ένα πράγμα, ότι δεν ζητούμε διαφοροποίηση μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και μικρομεσαίων. Το μόνο που ζητούμε είναι η οδηγία αυτή να επαναδιατυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έπειτα, για το ζήτημα του κυρίου Μάντερς και του κυρίου Ντεγιόγκ, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις εφόσον συμπεριλάβουμε τι σχέσει επιχειρήσεων προ επιχειρήσει, νομίζω ότι θα βελτιωθούν οι καταστάσει, ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Βεβαίω, πάντοτε θα υπάρχουν τομεί που δεν θα συμφωνούν. Αλλά αυτό ακριβώ είναι και το πρόβλημα με τι καθυστερήσει πληρωμών. Υπάρχουν σορευτικέ συνέπειε. Υπάρχει ένα φαινόμενο χιονοστιβάδα για όλου του τομεί που συμπεριλαμβάνονται. Το θέμα τώρα του αν θα θέλαμε οδηγία ή κανονισμό. Καλή πρόταση για κανονισμό, αλλά το πλεονέκτημα αυτή τη οδηγία είναι ότι σε κάθε περίπτωση μα ενδιαφέρει η εσωτερική αγορά. Οι μικρομεσαίε τη επιχειρήσει, ιδίω οι εξάγουσε, χρειάζονται σαφεί κανόνε. Σαφεί κανόνε που να είναι οι ίδιοι σε όλε τι χώρε. Ευχαριστώ για ένα λεπτό Έχω απλώ το χρόνο να απαντήσω στην κυρία Γκέπχαρντ. Βεβαίω τα δεδομένα που ανέφερα αφορούν το δημόσιο τομέα, τον υγειονομικό τομέα που έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στην πραγματικότητα, ο ιδιωτικό τομέα είναι πολύ πιο συγκατημένο στην Ιταλία και η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Οι πληρωμέ γίνονται πολύ πιο έγκαιρα, όχι πάντοτε απόλυτα εγκαίρος, 50% ε, γέρος και 35% με 30 μέρε καθυστέρηση. Όμως, οι ιδιωτικοί φορείς είναι οι πρώτοι που επιβαρύνονται από αυτή την κατάσταση, διότι είναι οι πρώτοι πελάτες ε, δημόσια δίκηση. Οπότε λαμβάνουν πληρωμέ με καθυστέρηση, δεν μπορούν να επενδύσουν περαιτέρω στην καινοτομία, την έρευνα, που για την υγεία είναι καθοριστική σημασία. Αυτή είναι η πραγματική στρέβλωση του ανταγωνισμού. Διότι και οι συνάδελφοι το ανέφεραν, το 25% των πτωχεύσεων επιχειρήσεων ιδιωτικών στην Ιταλία, βάσει των δεδομένων μα, οφείλονται στι καθυστερήσει πληρωμών. 25%. Φανταστείτε. Δεν ξέρω πόσε δημόσιε αρχέ, ε, επαρχίε, και νομή στην Ευρώπη πτωχεύουν λόγω καθυστέρησης πληρωμών των ιδιωτικών φορέων στις άλλες χώρες. Να ευχαριστήσω όλους μας τους ειδικού για τις πολύ καλές τους παρουσιάσεις, για τη διεξοδική απάντηση που έδωσαν σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Και τώρα θα ζητήσω την κυρία Μπρίγκμαν, τη Διευθύντρια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να απαντήσει θα τα καταφέρετε με αυτή τη σειρά των ερωτήσεων. Έτσι και αλλιώ θα ξανάρθετε στην Επιτροπή μα, αλλά θα σα δώσω πέντε λεπτά για να απαντήσετε τώρα. Και μετά θα καλέσω του δύο εισηγητέ μα να κάνουν κάποιε σύντομε καταληκτικέ παρεμβάσει. Ο κ. Μπαλτασάρα, η κυρία Βάιλερ. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν σε ένα τέταρτο. Ξεκινώ με την κυρία Μπρίγκμαν. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais, au nom de la Commission, euh, vous Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Επιτροπή, ευχαριστώ εσά και την κυρία Βάιλερ για αυτή την πρωτοβουλία. Euh, αυτή η συζήτηση έδειξε τον πλούτο των απόψεων, των αντιλήψεων όσον αφορά την υπερημερία στην Ευρώπη. Αλλά από την άλλη μεριά είδαμε και τι λύσεις μπορεί να προταθούν και να υιοθετηθούν από τον νομοθέτη. Ή κάποιοι από τους που έλαβαν λόγο μας ανέφεραν ότι αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ σημαντική, ούτω ώστε να βελτιωθεί η θέση των ΜΜΕ. Και ότι η πρότασή μας είναι πάρα πολύ βασική όσον αφορά το νομοθέτημα για τις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τις ΜΜΕ. Το έγγραφο εργασίας από την συγγήτρια και από όσους έλεγαν το λόγο εκφράζουν τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο και εγώ θέλω να σταθώ σε τρία σημεία. Αυτά τα οποία προσέξουμε περισσότερο κατά την διαδικασία της συναπόφασης. Συμφωνούμε ότι αυτά που σήμερα συζητήθηκαν είναι τα πιο σημαντικά που θα πρέπει οι συνομοθέτες να τα συζητήσουν και να αναζητήσουν κάποιες λύσεις δόκιμες. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά την διαφοροποιημένη αντιμετώπιση του κρατικού από τη μία και του ιδιωτικού τομέα από την άλλη. Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζει όντως διαφορετική μεταχείριση. Και είναι θεμετό αυτό το οποίο ετέθη. Ότι δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε να μην περιοριστεί, μην κολοβωθεί η ελευθερία των συμβάσεων. Κάθε φορά προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τις σχέσεις μιας επιχείρησης με το κράτος. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και πλευράς ε, δικαίου και του δευτερογενούς δικαίου. Έχουμε δεδομένα τη διάκριση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η ιδέα ελευθερία των συμβάσεων είναι κάτι το οποίο ελήφθη υπόψη όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τη σχετική οδηγία. Αυτό ορίστηκε ότι έχει θεσπιστεί για το κρατικό τομέα και όχι για τις επιχειρήσεις. Επομένως, να. Μπορούμε αυτή την τόσο θεμελιώδη αρχή να την λάβουμε υπόψη. Και να θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη όσον αφορά τη συμβάση που συνάπτονται μεταξύ δημόσιου και δυτικού τομέα. Και πάντοτε καταλήγουμε στο ότι αναδύονται προβλήματα και άρα θα πρέπει να καλύψουμε όλες αυτές τις ανησυχίες των ε, όσων έλαβαν τον λόγο. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις, συγκεκριμένα μέτρα. Όντω λοιπόν δικαιολογείται αυτή η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό κάτι να κάνουμε το ώστε να μην διασπαστεί, να μην διαταραχθεί η εσωτερική αγορά. Άλλωστε είναι αντίστοιχη και η νομική βάση. Η νομική βάση που αφορά την εσωτερική αγορά. Βεβαίω και υπάρχουν ε, διαφορετικέ ρυθμίσει όσον αφορά τι πλήρωμέ στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να μην εμποδιστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων. Άρα θα πρέπει να δούμε το ότι η περιμερία είναι ένας φραγμός όσον αφορά τη συμμετοχή των ε, επιχειρήσεων των διαφόρων χωρών ε, στους διαγωνισμούς και επομένως θα πρέπει να προστατεύσουμε την εσωτερική αγορά με κάποιες αυστηρές διατάξεις και έτσι να καταπολεμηθεί η υπερημέρεια. Είναι προηγούμενος κρίσιμη κατάσταση σε αυτόν τον τομέα. Και είναι ξεκάθαρο ότι συντρέχουν οι λόγοι Ούτω ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε την εύρεθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και έτσι δικαιολογείται η παρέμβασή μας. Και ένα σωρά άλλα επιχειρήματα έχουν ακουστεί, αλλά δεν να μην τα αναπτύξουμε τώρα στις λεπτομέρειές τους, αλλά εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει να γίνει διαφοροποιημένη αντιμετώπιση επίσης όσον αφορά το 3 ημέρα και όσον αφορά την αντίστοιχη επιβάρυνση ως κύρωση. Θεωρούμε ότι οι 30 μέρες ήδη ισχύουν ως προθεσμία σε πολλά κράτη-μέλη. Και άρα δεν μπορεί να ισχύει άλλο σε κάθε κράτος μέλος. Μεγάλη Βρετανία. Δέκα ημέρες προβλέπονται. 30 μέρες στη Γαλλία και στη Γερμανία ως πλήστον προβλέπεται προθεσμία κάτω από 30 μέρες. Άρα εμεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ισχύουν αυτές τις 30 μέρες, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας πυλώνας, είναι, είναι θεμέλιο για την πρότασή μας. Άλλωστε και το πρόγραμμα για την ανάκαμψη ορίζει ότι θα πρέπει οι κρατικές υπηρεσίες μέσα σε ένα μήνα να εξοφλούν τα χρέη τους. Επίσης, ε, υπάρχει προγραμματισμός για αυτό το 5%. Ελέγχει ε, ότι είναι ευθέρετο, ότι είναι δυσανάλογο. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Θέλουμε κάτι να θεσπιστεί. Κάτι το οποίο να αποτελεί κίνητρο για το κράτος να πληρώνει. Κύρωση, αλλά ρεαλιστική θα κάτσουμε και θα το μελετήσουμε σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί και εμείς και ο συνομοθέτης. Πρέπει το ίδιο το είπε και ο κύριος Μπαρνία. Κάτι αναλογικό, κάτι το προοδευτικό. Επίσης, υπήρξαν και άλλες προτάσεις προς αναζήτηση κάποιας ε, ισορροπημένης λύσης. Α, κάτι άλλο για τα κρατικά νοσοκομεία και τις σχετικές υπηρεσίες υγείας. Ξέρουμε, ξέρουμε ότι η διαχείριση των οικονομικών στα νοσοκομεία αυτά είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Ε, δεν υπάρχουν εισοδήματα σταθερά και είναι το θέμα εδώ επιδοτήσεων που καταβάλλονται οι ενισχύσεις ε, με καθυστέρηση και η διαχείριση των οικονομικών γίνονται από άλλες υπηρεσίες οπότε αυτή η κατάσταση δεν βοηθάει πάρα πολύ όσον αφορά τι τις ε, και την αποπληρωμή των χρεών αλλά το θέμα είναι είναι σωστό ο προμηθευτής να ε, πληρώνει αυτό την ύφη όσον αφορά αυτές τις, την κακή οργάνωση των, των ενισχύσεων των πληρωμών, ε, ε, τη διαχείριση των οικονομικών σε κάποια κράτη-μέλη. Αυτό να δούμε επομένω. Πώς θα γίνει προσαρμογή της χρηματοδότησης των νοσοκομείων στα όσα απαιτούνται να γίνουν. Έχουμε ένα σωρό καταγγελίες, ξέρετε, στην Κομισιόν όσον αφορά οι υπερημερίες. Και πάρα πολλέ από τις καταγγελίε αφορούν τέτοια. Κρατικά νοσοκομεία, Πρόεδρε, αυτά. Ελπίζω ότι... Α, α πέρασα τώρα, το πέρασα. Πάει. Ήμουν ιδιαίτερα γενναιόδωρο μαζί σα, γιατί αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ... ενδιαφέροντα. Και τώρα σχόλια από τους συζητητέ μας. Ο κύριος Ντεάντζελη και ο κύριος Μπαλτασάρε θα ήθελα να κάνουν σύντομα σχόλια. Και θα έχουμε και το χρονόμετρο για να μην χάνετε. Θα είμαι τηλεγραφικός, λέει ο κύριος Μπαλτασάρε. Το πεδίο της εφαρμογής όλα αυτά ανακαλύπτει και τους καταναλωτές. Θα πρέπει όμως το να προβλέψουμε κυρώσει για τους καταναλωτέ αυτή τη στιγμή μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Επίσης, θα πρέπει όσοι ασχολούνται με τον αντίκτυπο της οδηγίας αυτής να μην ξεχνούν τους εκπροσώπους των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει οι εκπρόσωποι των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης εφόσον παρουσιάζουν αρνητικά αποτελέσματα να μην ξεχνούμε ότι πολλέ φορέ αποτελούν τη μισή αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δύο μικρέ διευκρινήσει. Δεν αποκλείεται δυνατότητα να οριστούν διαφορετικοί χρόνοι προθεσμίες. Όμως θα πρέπει να περιορίσουμε τις δυνατότητες εξαιρέσεων για εξαιρετικές περιπτώσεις. Επιπλέον, προκειμένου να εξεύρουμε ισορροπία μεταξύ της δυνατότητας, της απαιτήσει των επιχειρήσεων και της συμβατικής ελευθερίας, θα πρέπει ίσως να προβλέψουμε μια προθεσμία ανώτερη των 30 ημερών, που θα ξεπερνιέται αρκετά εύκολα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ τάχιστος. Νομίζω ότι η συζήτηση που είχαμε ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική. Προέκυψαν διάφορα ζητήματα που θα πρέπει να εμβαθύνουμε για να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε το κείμενο της Επιτροπής. Αυτό είναι και ο στόχος μας. Επειδή η Οδηγία 35 του 2000 μεταξύ άλλων δεν επέλυσε τα προβλήματα, τα προβλήματα που σήμερα συζητούμε. Δύο σημεία τα οποία θεωρώ σοβαρότατα. Να περιορίσουμε και, και εγώ πιστεύω στο μέγιστο βαθμό θα έπρεπε τις δυνατότητες εξαιρέσεων και έπειτα για το χρόνο και το έγκαιρον της εφαρμογής των κανόνων. Για το ζήτημα των καταναλωτών, όπως είπατε, είναι ένα στοιχείο που, όπως προέκυψε από τη συζήτηση, θα πρέπει να το αξιολογήσουμε με προσοχή. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει δεσμευτικό όμως. Πιστεύω πάντως ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθεθεί εφόσον δεν γίνει απαραίτητη μελέτη για να επιληθούν τέτοια προβλήματα που τόσο πολύ πλήττουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με μια οδηγία που θα αφορά και τα 27 κρατημέλη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τους δύο συντάκτες μας, συγητές μας, για την συνεισφορά τους στην πρωινή μας αυτή συζήτηση. Ε, περιμένουμε με αγωνία τους καρπούς των διαβουλεύσεών μας, διαβουλεύσεών σας στις ερχόμενες συνεδριάσεις. Και τώρα ε, ο λόγος στην εισηγητρία κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι σκληρή δουλειά, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ακρόαση. Ακούσαμε όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις και θέλω να συγχαρώ την Κομισιόν εγώ παρά την κριτική που άκουσα σήμερα. Καλό είναι το ότι ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, ίσως λίγο κάποια χρόνια καθυστερημένα, αλλά είναι καλό το, το κάνει αυτό. Ακούσαμε και με τη δική σας αξιολόγηση αντικτύπων και με άλλες που διάβασα της Βρετανικής κυβέρνησης, διαφόρων οργανώσεων. Η καθυστέρηση των πληρωμών είναι υπαρκτό πρόβλημα εντός της Ένωσης και στα κράτη-μέλη. Και ειδικά τώρα είναι παράλογο γιατί έχουμε προγράμματα κρατικά ε, ενίσχυσης της οικονομίας και εδώ πέρα έχουμε κάτι πάει στην τελείω αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό το οποίο θα συζητήσουμε λοιπόν τι επόμενες εβδομάδες ε, με τους γεωδησηγητές είναι τρία θέματα. Πρώτον, πεδίο εφαρμογής. Εγώ θεωρώ ότι είχα δίκιο και οι δύο οδηγίες ε, περί δημοσίων προμηθειών θα συμπεριληφθούν και οι 17 και 18. Επίσης θεωρώ πως πράγματι θα συμπεριληφθούν και τα ιδιωτικά νοσοκομεία, όχι γιατί είπατε πως πληρώνουν ούτως ή άλλως την ώρα τους, αλλά γιατί δεν θέλουμε να έχουμε διακριτική μεταχείριση των δημοσίων νοσοκομείων. Και εκεί για το οποίο έχω κάποιες αμφιβολίες και δεν έλαβα οριστική απάντηση από την Κομισιόν είναι γιατί δεν συμπεριέλαβε τη συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Δεν μου το εξήγησαν μου είπατε γιατί μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο για τους Δήμους, αλλά ε, γιατί δεν συμπεριλάβατε τις επιχειρήσεις, το παρακάμψατε. Εγώ προσωπικά επίσης δεν θέλω να συμπεριληφθούν οι καταναλωτές. Δεν είναι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή επιτάπητος. Το δεύτερο που θα συζητήσουμε είναι οι ποινές Εάν, όπως είπε ο συνάδελφος από την Ολλανδία, να έχουμε ένα πιο έξυπνο σύστημα και αποτελεσματικότερο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποινές πρέπει να υπάρχουν χωρίς κυρώσεις ε, θα είναι και μη δεσμευτικό όπως η οδηγία του 2003 οι 30 ημέρες θα το δούμε αυτό πάρα πολύ σοβαρά. Αν διαβάσετε όμως, γιατί φαίνεται πάρα πολύ αυστηρό, αλλά αν διαβάσετε την οδηγία, υπάρχουν παραπάνω από μία τρύπες, παραθυράκια, υπάρχουν παραπάνω <coughs> από ένα σημείο στα οποία μπορεί να εξαιρεθεί κανείς. Βρίσκω εγώ πάρα πολλά. Εντάξει, μπορούμε να είμαστε, εάν θέλετε, ή κάπως γενναιόδοροι με τους Δήμους, αλλά πρέπει να είναι αιτιολογημένο τώρα για τις ε, εθνικές ιδιαιτερότητες. Ο κύριος Μάντερς ήθελε κανονισμό. Κοιτάξτε, αν συμπεριλάβουμε τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις συνήθειες, δεν θα γίνει τίποτα. Είναι κρίμα, γιατί υπήρχε στη Γερμανία είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι υπάρχει μία διαδικασία διαιτησίες πριν πριν καταλήξουν στο δικαστήριο και σε άλλες χώρες, σε μεγάλα συμβόλαια γίνεται μια προσπάθεια διετησίας πριν καταλήξουν στο δικαστήριο. Αυτό θα ήθελα να διατηρηθεί. Φοβάμαι πως βεβαίως με έναν κανονισμό δεν γίνεται κάτι τέτοιο, θα το δούμε όμως. Ναι, για τις ορθές πρακτικές θα κοιτάξουμε παντού, αλλά εμένα δεν μου επαρκεί, κυρία Μπρίνκμανς, το να πούμε ότι θα πάρουμε, δεν θα συμπεριλάβουμε το B2B γιατί έχουμε άλλα μέτρα όπως π.χ. μια εκστρατεία διαφημιστική. Δεν μου αρκεί. Εγώ θέλω κάτι δεσμευτικό. Γιατί ε, όλοι υποχρεωνόμαστε και πρέπει να έχουμε και καλά και να, να έχουμε και καλά παραδείγματα. Πλην του καλού Ολλανδικού παραδείγματος πρέπει να αναφέρουμε και το Βρετανικό που είναι πολύ ενδιαφέρον σύστημα αυτό το που κατονομάζουν επίσης και όσους είναι πάντα στην ώρα τους, τους διαφημίζουν. Και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά βεβαίως αυτό οφείλεται και στη διαφορετική κουλτούρα του καθενός και έτσι είναι, διαπιστώσαμε πως ε, κάποιες κουλτούρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κύριο λόγο στον Νότο, αλλά όχι μόνο αποκλειστικά, είναι ε, Χειρότερε και στου δύο τον και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό και άλλα συστήματα α πούμε τη Φιλανδίας είναι πληρώνουν στην ώρα τους και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Ε, πρέπει να το δούμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα. Είναι ενδιαφέρον γιατί δεν σημαίνει αυτομάτως πως ε, τα νέα κάπως φτωχότερα κράτη από την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη είναι κάπως χειρότερα. Δεν ισχύει αυτό αυτομάτως. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Για το χρονοδιάγραμμα να πω πως οπωσδήποτε μετά την ακρόαση αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να μην αναβάλουμε πλέον αυτή την οδηγία γιατί έχει καθυστερήσει ήδη καιρό, θα εργαστούμε γρήγορα, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε έντονα και με την Επιτροπή ε, Νομικών ε, υποθέσεων. Νομίζω ήδη στις 19 ε, θα μπορέσουμε να δώσουμε μία ε, έκθεση ήδη για μετάφραση και μετά να εχουμε δύο, τρεις, τέσσερις εβδομάδες με τους και ηγητές για να δούμε πολύ σοβαρά τι θα γίνει και με την Κομισιόν για να ξεκαθαρίσουμε τα ανοιχτά ζητήματα. Σας ευχαριστώ. well, I'd like to... Ο να ευχαριστήσω την Πάρμπαρα Βάιλερ ε, πραγματικά, ε, διότι ε, είχε την, την πρωτοβουλία για, για, για, αυτό που κάναμε. Ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η ακρόαση. Ευχαριστώ επίση για την ζωηρή συμμετοχή σα και ευχαριστούμε πάρα πολύ και του διερμηνεί μα παρεχώσαν χρόνο παραπάνω. Οπότε τώρα, εδώ τελειώνει η ακρόαση. Στι 3 η ώρα συνεχίζουμε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε όλο το απόγευμα και έχουμε και την εισήγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή ε, του κεκτημένου. Αφού θεσπίστηκαν κάποια πράγματα, είναι σημαντικό να δούμε την εφαρμογή τους πέρα στη συνεδρία